Uh, shall we start? Συνάδελφοι, μπορούμε να εργασίες μας. Δεν είμαστε πολύ πληθείς, αλλά είμαι σίγουρη ότι θα φτάνουν όλο και περισσότεροι με τις πτήσεις προς Βρυξέλλες Καταρχήν εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη. Υπάρχουν παρατηρήσεις. Φαίνεται πως όχι. Εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη όπως προτάθηκε. Αλφάνο, θα ήθελα να υποβάλω ένα ερώτημα ως προς την ημερήσια διάταξη. ως προς την ημερήσια διάταξη έλεγα, ως προς την ε, ψηφοφορία αύριο της έκθεσης Μακοβέη, όπως ξέρετε, η έκθεση Μακοβέη προβλέπεται για τις 3 και δυστυχώς συμπίπτει με τη συνεδρίαση της ΚΡΙΜ. Κάτι το οποίο δεν μπορεί να μετατεθεί, διότι θα έχουμε και την Επίτροπο Μάλστρεμ και ανταλλαγή απόψεων με βουλευτές από τα άλλα κράτη-μέλη. Γι' αυτό δεν μπορούμε να ακυρώσουμε ή να μεταθέσουμε την αυριανή συνεδρία. Επειδή ο εισηγητής, εγώ και άλλοι βρισκόμαστε και στη Λίμπε και στην Κρίμ, δεν θα θέλαμε... Μάλλον θα θέλαμε να δούμε τι μπορεί να γίνει ε, ως προς τις ψηφοφορίες το συζητήσαμε και με τους συντονιστές της ΚΡΙΜ. Ή μπορούμε τις αυριανές ψηφοφορίες της ΚΡΙΜ να τις μεταθέσουμε από τις 9 στις 9.30 για να μπορέσουμε αύριο εδώ να ψηφίσουμε την έκθεση Μακοβέη ή να ψηφίσουμε την έκθεση Μακοβέη στις 11 όταν λήξουν οι εργασίες της ΚΡΙΜ. Θα θέλαμε όμως να συμμετάσχουμε στις εργασίες και να μην ε, δημιουργήσουμε αρνητική εικόνα στους βουλευτές από τα άλλα κράτη και στην Επίτροπο Μάλστρεμ. Καταρχήν, επειδή, ο επειδή η συγγήτρια δεν είναι παρούσα, δεν ξέρω τι μπορούμε να κάνουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Έγιναν διαβουλεύσεις ε, για την πρόταση και δεν υπάρχει πλειοψηφία Κατανοώ το πρόβλημα, αλλά όπως και να διευθετήσετε την ψηφοφορία θα έχετε το ίδιο πρόβλημα, διότι συμπίπτουν οι επιτροπές. Εγώ έχω και άλλη επιτροπή στις ε, τρεις, γι' αυτό δεν νομίζω ότι αυτό μπορεί να επιληθεί. Είμαι πολύ επιφυλακτική, δεν θέλω να το αποφασίσω εν τη απουσία της εισηγήτριας. Θα ήθελα να παραμείνει ως έχει το θέμα. Madame la Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας ζητήσω να το ψηφίσουμε, να ψηφίσουμε από αυτού όπως πρότεινε η κυρία, Αλφάνο. Δηλαδή να μην πάρετε την απόφαση μόνοι σας. Πρόεδρος, όχι, δεν πήρα θέση. Είπα ότι, δεν, έχω την αίσθηση ότι δεν είναι καλό να πάρουμε οποιαδήποτε απόφαση ε, τη απουσία της ε, εισηγητρίας τότε ίσως να πούμε ότι θα το συζητήσουμε στο τέλος της συνεδρίασης έτσι ώστε να ρωτήσουμε την άποψη της συζητρίας, κυρία Ματιώ. Δηλαδή λέμε ότι αντί για τρεις το μεσημέρι να ψηφίσουμε στις 10 και 30 το πρωί και επομένως θα είναι ούτως ή άλλως παρόντες οι συνάδελφοι της ΛΥΜΠΕ γιατί θα είναι εδώ από τις 9 μέχρι τις 7.30 το απόγευμα. Ε, από την άλλη πλευρά, στην ε, Επιτροπή ΚΡΙΜ ε, θα έχουμε εκπροσώπου από 35 κοινοβούλια στα πλαίσια μιας ακρόασης μαζί με την Επίτροπο Μάλστρομ. Ε, ε, πρόκειται για μια ακρόαση σημαντική, ε, την έχουμε συζητήσει και συμφωνήσει πριν από πάρα πολύ καιρό και νομίζω ότι είναι και θέμα της εικόνας που θα δώσουμε. Δηλαδή να είναι 35 εκπρόσωποι Εθνικών Κοινοβουλίων και η κυρία Μάλστρομ η Επίτροπος και να μας περιμένει εμάς να τελειώσουμε την ψηφοφορία, δεν νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλό αυτό. Προτείνω λοιπόν να επανέλθουμε στο ζήτημα αυτό αργότερα το απόγευμα, έτσι ώστε να δούμε και το χρονοδιάγραμμα και να συζητήσουμε και με την εισηγήτρια. Συμφωνείτε πριν το πέρας της συνεδριάσεως, πριν τις μισή, να ξανασυζητήσουμε το θέμα. Να δούμε το πρόγραμμα λοιπόν, να ρωτήσουμε και την άποψη τη εισηγητρίας και να αποφασίσουμε. Ωραία θαύμα. Μία παρατήρηση όσον αφορά την συζήτηση για την προστασία των δεδομένων, κοινή συζήτηση που θα ξεκινήσει με τον κανονισμό και θα συνεχίσει με την οδηγία. Το επόμενο σημείο της σημερινής διάταξης είναι η παρουσίαση του κυρίου Γκέρουμα, ε, Διευθυντή του Οργανισμού Θεμελιδών Δικαιωμάτων, κατόπιν της επιστολής του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ε, του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 22 Απριλίου 2013 σχετικά με την πρόθεση του εν λόγω Διοικητικού Συμβουλίου να παρατείνει τη θητεία του Διευθυντού. Μπορείτε να περιμένετε ένα λεπτάκι. Ο κύριος Κέρωμα υπήρξε διευθυντής ε, του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων ΦΡΑ από το 2008. Ολοκληρώνεται η θητεία του σύντομα. Και επομένως θα σας δώσω αγαπητέ κύριε Κέρουμ 10 με 15 ε, λεπτά έτσι ώστε να αναφερθείτε στην θητεία σας και την υποψηφιότητά σας. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Είναι τιμή μου που βρίσκομαι σήμερα εδώ μετά από την ε, πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της, ε, του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων να παρατείνει την εντολή μου. Με μεγάλη μου χαρά επίσης καλωσόρισα την Επιτροπή Λίμπε στη Βιέννα πριν από μερικού μήνες στα κεντρικά μας γραφεία όπου είχαμε μια ε, πολύ καλή ανταλλαγή απόψεων, πολύ ζωντανή, πολύ αξιόλογη και πολλά άμεσα αποτελέσματα προέκυψαν από αυτές τις διαβουλεύσεις. Ελπίζω λοιπόν αυτό να συνεχιστεί και στο μέλλον. Πριν πέντε χρόνια, όταν βρισκόμουν σε αυτήν ακριβώ τη θέση, πριν από την οριστική απόφαση για, την, ε, για τον πρώτο διορισμό μου ω διευθυντή της ε, θέση αυτή, του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, υποσχέθηκα να δημιουργήσω μια ευρωπαϊκή αχτίδα προστασία για τα ανθρώπινα δικαιώματα και έναν καινοτόμο οργανισμό για τα θεμελιώδη δικαιώματα, καθώς και έναν οργανισμό όπου μπορεί κάποιος να απευθυνθεί για όλα τα ζητήματα ε, που τον αφορούν σχετικά με τα θεμελιώδη δικαιώματα. Μπορώ να πω τώρα ότι η αποστολή μου έχει εκπληρωθεί. Πρόσφατα μας έγινε εξωτερική αξιολόγηση, είχαμε μία έκθεση και οδηγηθήκαμε σε σημαντικά συμπεράσματα. Θα ήθελα να σας τονίσω ορισμένα από τα επιτεύγματα που καταφέραμε να έχουμε στα τελευταία πέντε χρόνια. Καταφέραμε να δημιουργήσουμε μία μοναδική συγκέντρωση δεδομένων, συγκριτικών δεδομένων για τα ανθρώπινα δικαιώματα και αναλυτικών στατιστικών στοιχείων. Όταν αρχίσαμε το έργο μας το 2007-2008 είχαμε ελάχιστα δεδομένα στη διάθεσή μας και αυτά τα δεδομένα δεν μπορούσαμε να τα συγκρίνουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στόχος μας ήταν να παρέχουμε τις αναγκαίες αποδείξεις έτσι ώστε να δημιουργήσουμε μια πολιτική βασισμένη σε στοιχεία στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Διεξάγαμε μελέτες κοινωνικές, οικονομικές ερωτηματολόγοι. Είχαμε πάνω από 100 εκθέσεις σε αυτά τα πέντε χρόνια που κάλυπταν ένα εύρος ε, θεμάτων σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτές οι εκθέσεις αποτελούν τη βάση των γνωμοδοτήσεων, των ενημερωτικών εκθέσεων και όλων των σχετικών εγγράφων που έχουν φτάσει στα χέρια σας και σας βοηθούν στο σημαντικό σας έργο, στο σημαντικό έργο αυτού του Κοινοβουλίου. Η συλλογή μας ε, αυτών των αναλυτικών συγκριτικών δεδομένων επιβεβαιώθηκε στην ε, εξωτερική αξιολόγηση εγκρίθηκε από πάνω από 300 ενδιαφερόμενους, μαζί ευρωβουλευτές, ε, μέλη ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και κράτη-μέλη και μέλη του Συμβουλίου. Το δεύτερο επίτευγμά μας τώρα, ο οργανισμός ΦΡΑ, έγινε ένας οργανισμός κεντρικός όπου, στον οποίο στρέφονται όλοι για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Συγκεντρώνει λοιπόν όλους τους ενδιαφερομένους σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και συγκεντρώνει και τις πολιτικές. Να σας δώσω ορισμένα παραδείγματα. Τον Ιούνιο, σε μερικές εβδομάδες δηλαδή από τώρα, θα ε, διεξάγουμε ένα συνέδριο που θα προωθεί το κράτος δικαίου. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που ο κύριο Σταβάρης από τη δική σας επιτροπή θα συμμετέχει στις συζητήσεις στην Βιέννη. Πριν από δύο εβδομάδες επίσης, ε, έλαβε χώρα η πλατφόρμα θεμελιωδών δικαιωμάτων στη Βιέννη. Συμμετείχαν όχι μόνο 250 μη κυβερνητικοί οργανισμοί από όλη την Ευρώπη, αλλά και τρεις συνάδελφοι, τρεις ευρωβουλευτές, αρκετοί υπάλληλοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εκπρόσωποι της Ιρλανδικής Προεδρίας, του Συμβουλίου της Ευρώπης, του ΩΣΑ, ορισμένους από τους κύριους εδώ δωρητές και σημαντικούς συμμετέχοντες. Ήταν λοιπόν ε, ένα πολύ σημαντικό φόρουμ για να συζητηθούν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η πλατφόρμα θεμελιωδών δικαιωμάτων έχει αποτελέσει πηγή έμπνευσης για παρόμοιες πλατφόρμες, για την ΕΑΣΟ, για παράδειγμα. Σε γενικέ γραμμέ μπορώ να πω ότι εμείς καταφέραμε να χτίσουμε έναν ισχυρό μηχανισμό συνεργασίας με άλλους ευρωπαϊκούς οργανισμούς, ιδιαίτερα με τις Ευρωπαϊκές Υπηρεσίες Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Συνεισφέραμε σημαντικά στην εφαρμογή της ε, στρατηγικής ε, ανθρωπινών δικαιωμάτων της ε, Frontex, αλλά και σε άλλους οργανισμούς. Για παράδειγμα, συντάξαμε μία κοινή έκθεση στην, με την υπηρεσία ελέγχου ασθενειών στην Στοκχόλμη. οι οποίοι συνειδητοποίησαν ότι στα πλαίσια των εργασιών τους ε, είχαν να κάνουν πολλά που αφορούσαν και τα ανθρώπινα δικαιώματα και έτσι λοιπόν η συνεισφορά μας ήταν σημαντική. Για παράδειγμα, όταν εμείς ε, διαπιστώνουμε ε, εμπόδια στην πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας για ορισμένες ομάδες, για τους Ρωμά, για παράδειγμα, αυτό αφορά και τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ε, υπηρεσίες υγείας. Τέλος, θα ήθελα να σας αναφέρω ότι πριν πέντε χρόνια όταν είχα έρθει εδώ, έλαβα από πολλού από εσά την ερώτηση του πώς θα συνεργαστούμε με το Συμβούλιο. Και εδώ θα σας παραπέμψω στην εξωτερική εξελόγηση που μας έγινε, στην οποία υπήρχε αρχικά ε, κριτική αντιμετώπιση, διότι ήμασταν ένας καινούριο οργανισμός. Αυτή όμω η αρχική κριτική αντιμετώπιση έχει μετατραπεί σε ενθουσιασμό για την συνεργασία μας. Επίση, να σας αναφέρω ότι το Δικαστήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έχει δημοσίευσει δύο έγγραφα. Το πρώτο ε, έχει να κάνει με τις διακρίσει, το οποίο έγινε ευρέως αποδεκτό και κυκλοφόρησε σε όλα τα κράτη-μέλη και ε, την επόμενη έκθεση για την μετανάστευση και τα ανθρώπινα δικαιώματα, η οποία θα δημοσιευθεί τον Ιούνιο. Συνεισφέρουμε στην δημιουργία προτύπων για πολλά θέματα, για, ε, τις, ε, για διάφορες ομάδες, τις γυναίκες, τους ΛΟΑΔ και άλλες επίσης. Αυτό που θέλω να πω εδώ είναι ότι είναι σημαντικό το γεγονός ότι εμεί καταφέραμε να δημιουργήσουμε αυτόν τον οργανισμό, πως καταφέραμε να δημιουργήσουμε στη Βιέννη αυτή την υπηρεσία με προσωπικό, το οποίο από 35 άτομα στην αρχή της εθιτείας μας έχει διευρυνθεί σε πάνω από 100 τώρα. έτοιμο να αντιμετωπίσει όλες τις προκλήσεις που υπάρχουν και που θα έρθουν. Χρησιμοποιούμε πολλά εργαλεία σχεδιασμών για πολλούς τομείς πολιτικής. Και επίσης συνεισφέρουμε στις αλλαγές και στις μεταρρυθμίσεις των παλαιών πολιτικών. Μπορώ να σας ε, διασφαλίσω σε αυτό το σημείο ότι εμείς έχουμε κάνει το καλύτερο δυνατόν για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που έχουν προκύψει όσο το δυνατόν γρήγορα και αποδοτικά. Ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων έχει γερούς μηχανισμούς σε λειτουργία. Το 2012 ο οργανισμός μας ήταν ε, ο μόνος ευρωπαϊκός οργανισμός που δεν είχε κανένα αρνητικό σχόλιο από το ηλεκτρικό συνέδριο. Και πολλές ευρωπαϊκές υπηρεσίες υιοθετούν ε, πάρα πολλά από τα προγράμματά μας και από τα εργαλεία σχεδιασμού που έχουμε δημιουργήσει. Πιστεύουμε πως μόνο με συμπαγείς εσωτερικές δομές θα καταφέρουμε να έχουμε τα καλά αποτελέσματα που είχαμε μέχρι τώρα. Θα ήθελα να σας πω τώρα δύο λόγια για το μέλλον, για το τι προτιθέμεθα να κάνουμε. Ένα από τα συμπεράσματα της εξωτερικής αξιολόγησης ήταν ότι ο οργανισμός μας θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ακόμα περισσότερο στα πλαίσια νομοθετικών εργασιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όπως γνωρίζετε όμως, ο οργανισμός μας παραμένει στην ε, διάθεση των ευρωπαϊκών οργανισμών κατόπιν αιτήματός τους. Πριν από μερικούς ε, μήνες στη Βιέννη, στην επίσκεψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διαπιστώθηκε ότι η δουλειά μας είναι πάρα πολύ σημαντική για τη δουλειά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και για, το, για τα έργα αυτής ε, της Επιτροπής. Καθ' όλη τη διάρκεια του 2012 επίσης συνεισφέραμε στο έργο αυτής της Επιτροπής συντάσσοντας γνωμοδοτήσεις για πολλές υποθέσεις κατόπιν δικού σας αιτήματο. Πώς μπορούμε τώρα να προχωρήσουμε ακόμα πιο πέρα όσα έχουν ήδη γίνει. Εδώ θα πρότεινα να δημιουργήσουμε μια τακτική ανταλλαγή μεταξύ ημών και ημών η οποία θα ανταποκρίνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις ανάγκες σας. Πιστεύω πάντως πως αυτή η τακτική ανταλλαγή απόψεων θα βοηθήσει πάρα πολύ και εμάς και εσάς. Επίσης, επιθυμούμε να ενισχύσουμε τη συνεργασία με ορισμένα κράτη-μέλη και με όλα μάλλον τα κράτη-μέλη για ορισμένα θέματα. Όμως, οι πόροι είναι Περιορισμένοι, όπως γνωρίζετε. Υπάρχουν όμως ορισμένες έξυπνες μέθοδοι που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Πειραματιστήκαμε δημιουργώντας μικρές ομάδες εργασίας με τα κράτη-μέλη, για παράδειγμα στην αντιμετώπιση του ζητήματος των Ρωμά και του πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τους ε, δείκτες και τα στατιστικά στοιχεία για τις εθνικές στρατηγικές, για την ε, παράνομη μετανάστευση. Επίσης είχαμε συζητήσεις σε μικρές ομάδες με τους ε, υπουργούς εσωτερικών των κρατών μελών, καθώς επίσης και για τα εγκλήματα μίσους. Τέλος, αντικείμενο των συζητήσεών μας ήταν και η μεταρρύθμιση του οργανισμού. Διαπιστώθηκε η ανάγκη λισαβονοποίησης του κανονισμού, έτσι ώστε ο Οργανισμός Μελιωδών Δικαιωμάτων να γίνει ένας πλήρης ευρωπαϊκός οργανισμός που να καλύπτει όλους τους πυλώνες. Ελπίζω πραγματικά η Χάρτα των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων αποτελέσει τον σκελετό και τη ραχοκοκαλιά, αν θέλετε, των εργασιών μας. Τέλος, να σας πω, να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία που μου δώσατε να συνεισφέρω στην δημιουργία του πρώτου θεσμικού οργάνου του 21ου αιώνα για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Με μεγάλη μου χαρά είδα ότι πολλοί συνάδελφοι στη Βιέννη είχαν τη διάθεση να πάνε ένα βήμα παραπέρα, να δημιουργήσουν αυτόν τον μοναδικό οργανισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και επίσης θα ήθελα να πάρω αυτή την ευκαιρία να ευχαριστήσω εσάς, την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ, για την στήριξη και την επικοδομητική κριτική που μας δώσατε τα τελευταία χρόνια. Ευχαριστώ λοιπόν πολύ για την συνεισφορά σας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κιουέρουμ. Έχω τέσσερις συναδέλφους που θέλουν να πάρουν το λόγο. Κυρία Γκιόνς, κύριος Παλαιολόγος, κυρία Ντάνουκα. Υπάρχει κάποιος άλλος? Θα ήθελα να σας ζητήσω παρακαλώ να είστε σύντομοι, διότι μας μένουν 10 λεπτά. Κυρία Γκιόντς. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη πράγματι. Καταρχήν θα ήθελα να αναφέρω ότι, το, ότι βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη περίοδο για τον οργανισμό γιατί αυτό μας ενδιαφέρει είναι να δούμε ποια θα είναι, ποιο θα είναι το ρυθμιστικό πλαίσιο λειτουργίας και νομίζω ότι η περίοδος λειτουργίας ήταν πολύ αποτελεσματική. Έχω εκτιμήσει την εργασία σας, εργασία σας με μήκυο και είδα κάτι το σπάνιο για τα θεσμικά όργανα δηλαδή εταιρικέ σχέσεις επικοινωνίας με τις ΜΚΟ. Το κατανοώ αυτό γιατί είναι ύψη της σημασίας για την εργασία σας να έχετε και input και ε, υπάλληλου επιτόπου που να εργάζονται να εργάζονται επιτοπίως για την πρόθεση των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Αναφερθήκατε όμως σε ορισμένες πτυχές που συζητήσαμε εδώ αρκετές φορές. Είναι περιοριστική η ερμηνεία της χάρτας και ο τρόπος εργασίας σας επ' αυτής. Μπορείτε να διευρύνετε το πεδίο εφαρμογής αν συνεχίσετε με την εντολή σας έτσι ώστε να έχετε μία συνεχή εποπτεία του κράτους δικαίου και των κανόνων δημοκρατίας γιατί είναι μια απόλυτη αναγκαιότητα για να επιληθεί το δίλημα της Κοπενχάγης. Ένα άλλο ερώτημα. Πώς θα προωθήσετε το, το πολιτισμικό υπόβαθρο των θεμελιωδών δικαιωμάτων στα κράτη-μέλη. Ρομέρο Λόπες. Ευχαριστώ κύριε Διευθυντά του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Θα ήθελα να σας μιλήσω για την δουλεμπορία των γυναικών και την βία κατά των γυναικών. Η Επίτροπος Ρέντινγκ ανέθεσε στην Επιτροπή Βίλνιους μία μελέτη για τις γυναίκες στα πλαίσια θέσπισης ενός παρατηρητηρίου για τη βία κατά των γυναικών στην οικογενειακή αιστεία και εκτός η οικογενειακής ε, αιστείας, διότι η δουλεμπορία των γυναικών και η κακομεταχείρισή τους σχετίζεται με ευρύτερα δίκτυα στην Ευρώπη. Τι δυνατότητες ε, έχει ο οργανισμός για να ζητήσει από τις κυβερνήσεις αυτά τα δεδομένα που ζητούμε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δηλαδή στατιστικές της Eurostat. Ξέρουμε ότι και οι κυβερνήσεις δεν θέλουν να μας χωρίσουν αυτά τα στοιχεία. Θα ήταν όμως σκόπιμο να μάθουμε το πεδίο αυτό του φαινομένου σε σχέση με την βία των γυναικών, την κακομεταχείριση και την εμπορία τους. Μπορείτε να κάνετε κάτι η κυρία Αντωνούκα. Ευχαριστώ. Απλώς ε, ορισμένες δηλώσεις θα ήθελα να κάνω εντάχει. Ήμουνα εισηγήτρια για το ε, πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Ξέρετε ότι υπάρχουν προβλήματα με το Συμβούλιο, έτσι φαινόταν, αλλά τώρα έχει επιληθεί το θέμα και θα ήθελα να συγχαρώ την ΦΡΑ για το πεδίο εφαρμογής και τη λειτουργία της. Δεν είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι με τη λισαβονοποίηση όπως την αναφέρατε. Σας εύχομαι κάθε επιτυχία και σε εσά και στην Επιτροπή, Επιτροπή ΛΥΜΠΕ και βεβαίως θα πρέπει να τροποποιήσουμε το βασικό κανονισμό. Αυτό είναι, αυτό το βασικό μας μέλημα. Θα τα καταφέρουμε και υποστηρίζω την παράταση της θητείας του κυρίου Κερόμ γιατί ήταν αποτελεσματική η εργασία βεβαίως με ορισμένους περιορισμούς που επιβάλλονται από τον κανονισμό. Το ξέρουμε πώς μπορείτε να δουλέψετε κάτω από αυτές τις συνθήκες. Ευχαριστούμε η κυρία Γιάροκα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και την εργασία του οργανισμού σας τα τελευταία χρόνια. Πολλά νέα θέματα έχουν θυγεί εξαιτίας της δέσμευσής σας και το θέμα των Ρωμά ήταν ένα από αυτά μέσα στα πλαίσια της στρατηγικής στα τρία θεσμικά όργανα. Μας υποστηρίξατε, ε, λοιπόν, και θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Θα ήθελα να υποστηρίξετε τη θέση της Επιτροπής ε, ΦΑΜ έτσι ώστε να έχει λεπτομεριακή στοιχεία για ε, την έκθεση αξιολόγηση του Συμβουλίου, του Κοινοβουλίου, με Τους επόμενους μήνες θα παρευρεθούμε στην Κροατία για να διαπιστώσουμε την κατάσταση και σας, ε, θα θέλαμε να μας δώσετε υλικό πριν μεταβούμε εκεί. Η εκπαίδευση, η κατάρτιση και η στέγαση έχουν μεγάλη σημασία και ασχολείστε και με θέματα εμπορίας και γνωρίζουμε ότι έχετε στοιχεία ήδη από το 2011. Αυτά τα στοιχεία θα ήταν πολύ χρήσιμα για μας για τη μεγάλη έκθεση της Επιτροπής ΦΑΜ. Γιατί θα προετοιμάσουμε και την ημέρα της γυναίκας ε, για το 2014. Θα θέλαμε να δώσετε προτεραιότητα σε αυτό το θέμα. Δηλαδή να έχουμε μία εισήγηση νωρίτερα. Και σας ευχαριστώ για τη δέσμευσή σας Προσδοκώ να συνεργαστούμε και στο μέλλον. Δεν ξέρω κατά πόσο κάποιος άλλος ε, ζητά τον λόγο, φαίνεται πως όχι. Συνεπώς ε, θα υποβάλω κι εγώ μία τελική ερώτηση. Θα ήθελα και εγώ να σας συγχαρώ με τη σειρά μου για την εξαιρετική σας εργασία τα τελευταία χρόνια, πέντε χρόνια. Ε, υποβάλλατε μερικές εκθέσεις και θα ε, υποβάλλετε και μία έκθεση την επόμενη εβδομάδα για την ομοφιλοφοβία. Αλλά το ερώτημά μου είναι πολιτικής ε, υφής για το ρόλο του οργανισμού και τον ηγετικό σας ρόλο, γιατί είστε και ο πρώτος διευθυντής και προσπαθείτε να διαμορφώσετε το ρόλο του οργανισμού. Η Kinga Gens υπόβαλε μία παρόμοια ερώτηση. Ο οργανισμός ε, δικαιωμάτων, θεμελιωδών δικαιωμάτων, πώς πρέπει να λειτουργεί ως μια επιτροπή μελετών ή ως watchdog. Νομίζω ότι θα πρέπει να δεχτούμε και να δούμε αν πρόκειται για, μία, για ένα οργανισμό εκπόνησης μελετών, τότε θα πρέπει να αλλάξουν οι συνθήκες και να γίνει μία λησαγωνοποίηση, διότι θεωρώ ότι ένας οργανισμός θα πρέπει να είναι παρατηρητήριο και επόπτης. Ε, γιατί αν, κάνετε το, αν επιτελέσετε το ρόλο σας σωστά, όλα τα κράτη σας μισούν. Έμπρακτα, τι θα γίνει. Έχετε εκπονήσει μελέτες με εξαιρετικές συστάσεις αλλά τι βλέπουμε, λιγότερες ε, παραβιάσεις θεμελιωδών δικαιωμάτων στα κράτη-μέλη, όχι. Απελάβουν Ρωμά, ε, εκφοβίζουν τις γυναίκες, φημώνουν τον τύπο, προωθούν την ομοφιλοφοβία, άρα πώς θα κινηθείτε την επόμενη πενταετία. Υπάρχει και ένα επιστημονικό συμβούλιο και έχω την εντύπωση ότι υπάρχουν ε, άνθρωποι ή οργανώσεις που προβάλλουν απόψεις περί δημοκρατίας, αλλά δεν ε, κάνουν τίποτα άλλο παραβλέπουν τα θεμελιώδη δικαιώματα. Δηλαδή, τι κάνετε τη στιγμή που μία οργάνωση στρέφεται κατά των ομοφιλοφίλων, λεσβιών και ούτω καθεξής, τι κάνετε, πώς τους διώκετε, για να το θέσω έτσι. Δεν είσαστε μόνο ένας πολιτικός οργανισμός, υπάρχει και η διοικητική πτυχή. Μιλήσατε για προσωπικό και είπατε ότι ένα μέρος του προσωπικού δεν είναι ικανοποιημένο από τις μεθόδους εργασίας. Πρόκειται και για κάτι περισσότερο. Πολλοί άχθησαν ενώπιον της δικαιοσύνης, αλλά πολλές φορές η προσφυγή δεν ήταν έκνομη. Επειδή λοιπόν υπάρχει, υπάρχει αυτή η φημολογία θα πρέπει να δούμε κατά πόσο μπορούμε να μειώσουμε αυτούς τους φόβους. Τι έχει γίνει με τους καταδότες, πώς μπορείτε να αποκαταστήσετε τα πράγματα και να μας πείτε κατά πόσο υπάρχουν πρόσωπα που αποτέλεσαν αντικείμενο οχλήσεων ή παρενοχλήσεων. Νομίζω ότι αυτό το πολιτισμικό υπόβαθρο θα πρέπει να ε, διαγραφεί ή να απαλληλθεί. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ για τα ερωτήματα. Θα τις απαντήσω μία-μία. Χαίρομαι που σε ξαναβλέπω. Είχαμε συνδυθεί και στην πλατφόρμα των θεμελιωδών δικαιωμάτων και εκτιμήσαμε ιδιαίτερως και εμείς ε, αλλά και η κοινωνία των πολιτών την παρουσία των ε, ε, ευρωβουλευτών στην πλατφόρμα αυτή. Είχαμε και αξιωματούχους επιτροπής και εκπροσώπους της Προεδρίας και του Κοινοβουλίου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που είχαν τη δυνατότητα να συναντηθούν με εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών και να συζητήσουν για θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Uh, which cut πολλά και διαφορετικά ζητήματα ε, και αυτό το εκτιμήσαμε όλοι πάρα πολύ και ευελπιστούμε ότι θα συνεχιστεί αυτή η συνεργασία. Όσον αφορά την συστελτική ερμηνεία της ε, χάρτας ε, και του κανονισμού, πρέπει να πω ότι εγώ πήρα θέση από την αρχή και και όταν άρχισα να δουλεύω στην, ε, ε, ε, στον οργανισμό, αποφάσισα ότι θα πρέπει και ως νομικός βεβαίως να παραμείνω εντός των ορίων του κανονισμού έχοντας βεβαίως καλά αναλύσει τον λόγο κανονισμό ε, ε, και όπως είπατε και εσείς κυρία Πρόεδρε, μια και ήμουνα ο πρώτος υπεύθυνος αυτού του οργανισμού από την ίδρυσή του, ε, έπρεπε να ανοιχνεύσω λίγο το έδαφος, να δω τι μπορεί να κάνει, τι πρέπει να κάνει, με ποιο τρόπο μπορεί ο οφείλει να συνεργαστεί με υφιστάμενους οργανισμούς κλπ. Γιατί ξέρετε ότι στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων υπάρχουν πολλοί πρωταγωνιστές και σε εθνικό και σε υπερεθνικό επίπεδο ενώ έπρεπε να αναρωτηθούμε εξ αρχής ε, πού μπορούμε να προωθήσουμε τη δουλειά μας. Έχουμε ε, δημιουργήσει λοιπόν και έχουμε καταλάβει ε, έναν αρκετά σημαντικό χώρο γιατί υπάρχει μια σημαντική κόχη της αγοράς την οποία εντός αγωγικών της αγοράς την οποία μπορούμε να καλύψουμε. Η κύρια συζήτηση ε, σε αυτήν την ε, πρώτη θητεία ήταν η άμεση ελευθερία. Τώρα ε, θέλουμε βεβαίως να εξελίξουμε την συζήτηση αυτή. Ήδη συζητούμε με την ε, Κομισιόν για τις ε, διάφορες υφιστάμενες ε, δυνατότητες. Δοκιμάζουμε το έδαφος λοιπόν, βλέπουμε τι νέες πιθανότητες έχουμε και δυνατότητες, αλλά βεβαίως κάνουμε και δουλειά ανά περίπτωση. Γι' αυτό λοιπόν συνεδριάζουμε συχνά με τους συντονιστές για να βλέπουμε και πιο συγκεκριμένα θέματα. Αναφερθήκατε ειδικά και στο δίλημα της Κοπενχάγης, ε, το οποίο έχει πολλαπλά συζητηθεί. Όπως είπα και στην αρχή, έχουμε αυτό το συμπόσιο ε, ή σεμινάριο το οποίο θα διοργανωθεί τον ε, Ιούνιο και όπου θα έχουμε εκπροσώπους και από την Κομισιόν και από το Κοινοβούλιο ε, για να ε, δούμε ακριβώς ε, ποια, ποιοι είναι οι δείκτες που πρέπει να βλέπουμε, ποιοι είναι οι δείκτες οι οποίοι θα μας δείχνουν ότι τα πράγματα προχωρούν προς τη σωστή κατεύθυνση και ότι το κράτος δικαίου και ο νόμος εφαρμόζονται ορθά έχουμε ας πούμε δείκτες όπως είναι η ανεξαρτησία του δικαστικού τομέα ή η ανεξαρτησία άλλων οργανισμών ε, ή άλλων εξουσιών, ε, η αναφορά ε, εγκλημάτων μίσους. Όλα, όλοι αυτοί οι δείκτες οι οποίοι μας οδηγούν σε προώθηση των δημοκρατικών αρχών. Και βεβαίως... Στον οργανισμό μπορούμε ε, και βάσει της εντολής που έχουμε να προχωρήσουμε στην, στην κατεύθυνση αυτή. Βεβαίως βλέπουμε και ε, ε, τους επαγγελματίες των διαφόρων τομέων με τους οποίους μπορούμε να συνεργαστούμε. Αλλά ξέρετε υπάρχουν και κάποιοι περιορισμοί σχετικά με το πώς μπορούμε να επιτύχουμε σωστή επαφή με το ευρύ κοινό. Εμείς ε, ερχόμαστε, προτιμούμε να δουλεύουμε ε, με τους κοινωνικούς λειτουργούς, ε, με εργαζόμενους σε κοινωνικούς φορείς. Κυρία Λόπες, σχετικά με την ενδοοικογενειακή βία και την παρακολούθηση αυτής. Ξέρετε ότι έχουμε ξεκινήσει τη μεγαλύτερη μέχρι τώρα ε, επιθεώρηση έρευνα για το θέμα αυτό ε, στην Ευρώπη όπου βλέπουμε ενδοοικογενειακή βία, βία κατά των γυναικών, ε, βία ή παρενόχληση ή παρακολούθηση γυναικών στον χώρο εργασίας τους κτλ θέλουμε και μέσω συναδρίων αλλά και μέσω άμεσης επαφής με τις, χώρε μέλη ε, να συζητούμε έτσι ώστε να βρίσκουμε τα άμεσα και από τα μέτρα τα οποία μπορούν να λαμβάνονται. Υπάρχουν χώρες οι οποίες μας βοηθούν γιατί έχουν ε, πολλά και λεπτομερή στοιχεία αλλά αντίστοιχα υπάρχουν και χώρες οι οποίες δεν έχουν σχεδόν κανένα στοιχείο από αυτού ε, του ζητήματος και επομένως εκεί πρέπει να ε, κάνουμε τις δικές μας έρευνες. Αυτό που θέλουμε και εδώ είναι να καθορίσουμε μία σειρά δικτών έτσι ώστε να ε, ε, επιβάλλουμε ε, την ελάχιστη συλλογή στοιχείων και δεδομένων για κάθε χώρα. Όσον αφορά το τράφικινγκ, την εμπορία ανθρώπων, μιλάμε και με τον συντονιστή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το θέμα αυτό και προσπαθούμε να συντονίζουμε τις προσπάθειές μας. Ευχαριστώ την Στανούκα για, ε, ε, για τα καλά λόγια. Παρατήρηση ε, για τους Ρωμά. Θα επαναφέρω την πρόταση να προωθηθεί το θέμα των γυναικών Ρωμά. Αλλά επιτρέψτε μου, μια και έχω την ευκαιρία να πω ότι μία από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε, και εδώ απαντώ εν μέρη και στα δική σας ερώτηση, είναι ότι έχουμε ένα πάρα πολύ μεγάλο αριθμό στοιχείων πολλά δεδομένα λοιπόν τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πολλαπλές περιπτώσεις και σε πολλές ε, χώρες μέλη. Δεν έχουμε όμως πάντα και όλους τους πόρους έτσι ώστε σε βάθος να αναλύσουμε τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας Προσπαθούμε να κάνουμε εταιρικέ σχέσεις με άλλους οργανισμούς, με πανεπιστήμια, ακαδημαϊκούς φορείς κτλ. έτσι ώστε να μπορέσουμε ε, σύντομα και σε συγκεκριμένα χρονικά περιθώρια να επανέλθουμε ε, σε εσά και να δώσουμε συγκεκριμένες απαντήσεις. Όσον αφορά τον ρόλο του οργανισμού, I think we are, I think in between. Uh, και όσον αφορά τη θέση του Προέδρου και ε, εσείς κάνατε το σχετικό ερώτημα κυρία Πρόεδρε. Πρέπει να σας πω ότι δεν είμαστε μονάχα ε, οργανισμός ο οποίος ασχολείται και προμηθεύει, παρέχει μελέτες. Θέλουμε ε, να βρίσκουμε τρόπους χρήσης των στοιχείων και των δεδομένων αυτών. Να δούμε δηλαδή πώς μπορούμε να βρούμε άλλωστε και τα στοιχεία αυτά τα οποία θα κάνουν τη διαφορά που θα επιτρέψουν είτε στους εξωματούχους της Κομισιόν είτε ε, στα κράτη-μέλη να τους βοηθήσουν λέω να βελτιώσουν την κατάσταση σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Είναι γεγονός ίσως ότι ξοδέψαμε πολλούς πόρους και καταβάλαμε μεγάλες προσπάθειες έτσι ώστε να οικοδομήσουμε αυτό το πλαίσιο γνώσεων, τεχνογνωσίας, δυνατοτήτων ε, ε, έτσι ώστε να μπορούμε να κάνουμε ε, μελέτες σαν αυτήν που αναφέρατε για τους ΛΟΑΔ. Είχαμε ένα πάρα πολύ σημαντικό αριθμό απαντήσεων όσον αφορά την έρευνα για την ΛΟΑΔ, όπως επίσης και για την βία κατά των γυναικών. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτά, αυτά τα στοιχεία απορροφούν ε, μεγάλο μέρος του δυναμικού μας και των προσπαθειών μας αλλά παρόλα αυτά πρέπει να σας πω ότι για αυτά τα θέματα τουλάχιστον ε, βάσει των στοιχείων που έχουμε παράσχει εμείς ε, τα κράτη-μέλη πήραν συγκεκριμένα μέτρα. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να παρέχουμε στοιχεία τα οποία είναι ενδιαφέροντα για σας ε, και μάλιστα να τα παρέχουμε με τρόπο τέτοιο που να σας βοηθούν να, τα, να εφαρμόσετε μέτρα άμεσα. Ε, νομίζω ότι είναι γεγονός ότι αυτό που χρειάζεστε περισσότερο είναι αυτό που είχαμε κάνει ε, με τα δελτία δεδομένων, τα fact sheets ε, για τα εγκλήματα μίσους ας πούμε. Ε, είναι αλήθεια ότι δεν θέλουμε μία μικρή πλατφόρμα ε, δικαιωμάτων, θέλουμε μία ε, ευρεία πλατφόρμα θεμελιωδών δικαιωμάτων σε συνεργασία με όλους τους με όλους τους αντίστοιχους αρμόδιους φορείς. Επίσης, ξέρετε, ίσως ότι έχουμε καταρτήσει, ε, μάλλον έχουμε δουλέψει και πάνω ε, στις σχέσεις ε, με τους άλλους οργανισμούς και μάλιστα έχουμε αποκλείσει έναν οργανισμό που ασχολείται με τα ανθρώπινα δικαιώματα λόγω μη σεβασμού των αρχών μας. Και τώρα προχωράμε ακόμα περισσότερο στην κατεύθυνση αυτή. Επαγρυπνούμε λοιπόν. Θέλουμε βεβαίως όσο περισσότεροι φορείς ε, να συνεργάζονται μαζί μας, με την προϋπόθεση όμως ότι σέβονται τον διάλογο. Όσον αφορά τους whistleblowers, ε, εδώ μαζί με το Διοικητικό ε, Συμβούλιο προσπαθούμε να προωθήσουμε τις υποθέσεις. Δεν έχουν ολοκληρωθεί όλες. Υπάρχει ακόμα μία ε, υπόθεση η οποία ε, θα συζητήθηκε στις 2 Μαΐου ενώπιον του δικαστηρίου. Αναμένουμε λοιπόν την εκκρεμούσα δικαστική απόφαση. Ε, πάντως γενικά να πω ότι η πρόοδος είναι πάρα πολύ μεγάλη. Ευχαριστώ. Μάλιστα αυτό ολοκληρώνει και αυτό το σημείο της μερικής διάταξης. Έχουμε χάσει λίγο χρόνο. Θα προχωρήσουμε αμέσως στο επόμενο σημείο. Η δέσμευση και η δίμευση των προϊόντων εγκλήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η έκθεση Μακοβέη. Έχουμε περίπου μία ώρα για αυτό το σημείο. Και από ό,τι βλέπω δεν έχουμε σχόλια. Έχουμε λοιπόν μια παρουσίαση της νομικής υπηρεσίας του Κοινοβουλίου για την οδηγία που έχει προταθεί για την δέσμευση και δίμευση που έχει ζητηθεί από αυτήν εδώ την Επιτροπή. Θα επανέλθουμε στο θέμα της ψηφοφορίας μετά από διαβουλεύσεις. Τώρα η νομική υπηρεσία θα μας διευκρινίσει τη θέση της όσον αφορά τη νομική βάση και το πιθανό πεδίο εφαρμογής του οργάνου που θα καλύπτει τις ε, δημεύσεις, τη νομική βάση, καθώς και την επαναχρησιμοποίηση των περιουσιακών στοιχείων. Θα ήθελα να δώσω το λόγο τώρα στον κύριο Καϊόλα καταρχάς από την νομική υπηρεσία του Κοινοβουλίου. Έπειτα, το λόγο θα πάρει η συγγήτρια, σκιώδη συγγητή και όποιο άλλο βουλευτή θα ήθελε να συμμετάσχει. Κύριε Καϊόλα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα σας παρουσιάσω εν συντομία τι απαντήσει ε, στις τέσσερις ερωτήσεις που τέθηκαν στην νομική υπηρεσία του Κοινοβουλίου για την ε, προτινόμενη οδηγία δίμευσης και δέσμευση περιουσιακών στοιχείων προϊόντων εγκλήματο. Τώρα, στην πρώτη, όσον αφορά την πρώτη ερώτηση για τι πιθανότητες αποδεικτικών στοιχείων και τη νομική του βάση. Στάθμιση πιθανότητων, λοιπόν. θεωρούμε τα άρθρα 82 και 83 της συνθήκη σε σωστή νομική βάση. Ποινικές, καταρχάς οι ποινικέ διαδικασίες, οι ποινέ θα πρέπει να έχουν χαρακτηριστικά ποινών που δίδονται σε ποινικά αδικήματα και στις, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις διασυνοριακών εγκλημάτων παραπέμπουμε στο άρθρο 83 παράγραφος 1 όσον αφορά την δέσμευση μη βασιζόμενη σε καταδίκη. Θέλουμε μια ξεκάθαρη σύνδεση με την εγκληματική διαδικασία. Μέχρι τώρα η βάση μας ήταν η ε, ε, συνεργασία όσον αφορά την, τις δικαστικές διαδικασίες. Λέμε λοιπόν ότι ε, οι διαδικασίες οι οποίες αφορούν συγκεκριμένο άτομο και που ενδεχομένως οδηγούν σε ποινική καταδίκη βάσει της περιπτώσεως όπου υπάρχει ποινική καταδικαστική απόφαση σε αυτή την περίπτωση ε, θεωρούμε ότι η επιλογή της ε, στάθμισης πιθανότητων μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα. Ε, διότι ενδεχομένως θα δημιουργηθούν, θα εγερθούν ζητήματα όσον αφορά την αρχή της αναλογικότητας και της επικουρικότητας έτσι όπως αυτές οι αρχές αναφέρονται στις ε, τα, συνθήκες. Βάσει του 65.1 της συνθήκης λειτουργίας αναφέρεται ότι στον τομέα της ελευθερίας και της ε, ελεύθερης κυκλοφορίας θα πρέπει να γίνονται σεβαστές οι αρχές των κρατών Άλλωστε αυτό αναφέρεται και στο άρθρο 82 που αποτελεί την, μία από τις δύο παρούσες νομικές βάσεις για αυτήν την οδηγία. Ε, μία διαφορετική αντιμετώπιση θα μπορούσε να θεωρηθεί υπερβολική, ανά, ε, υπερβολική ανάμιξη ε, ε, όσον αφορά την ικανότητα απόδειξης ε, και επομένως να αντιτίθεται στην αρχή της επικουρικότητας και της αναλογικότητας σύμφωνα με το άρθρο 67. Ε, στην περίπτωση της ε, ε, συνεργασίας, η έκδοση αποφάσεων δίμευσης προϋποθέτει εν γέννη ποινική καταδικαστική απόφαση σε ορισμένες περιπτώσεις αυτό μπορεί να σημαίνει ότι το βάρος της, απόφα... απόδειξης θα πρέπει να είναι ικανόν ε, έτσι ώστε να ευθυγραμμίζεται με τις ε, ποινικέ αρχές. Ε, σε διαφορετική περίπτωση η χρήση της στάθμισης πιθανοτήτων δεν καλύπτεται από τις νομικές βάσεις των άρθρων 82 και 83. Τώρα, η εφαρμογή αυτής της βάσης σε δήμευση που δεν βασίζεται σε έκδοση απόφασης. Αυτό προβλέπεται στην παρούσα ε, οδηγία με την προϋπόθεση πάντως ότι η, δέσμευση, η δήμευση συγγνώμη, ε, ε, θεωρείται κύρωση βάση καταδικαστικής απόφασης. σε, σε αυτή την περίπτωση όμως το άρθρο 83 δεν μπορεί να αποτελέσει την σωστή νομική βάση, διότι, δεν, ε, ε, ε, διότι στην προκείμενη περίπτωση αυτό δεν εμπίπτει εις το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας. Σε αυτήν την περίπτωση έχουμε μετάθεση και εφαρμογή άρθρων της, του, αστικής, του αστικού κώδικα. Τώρα, ε, η έκδοση απόφασης δίμευσης ε, η οποία δεν βασίζεται σε ποινική καταδικαστική απόφαση ε, προϋποθέτει συγκεκριμένες διαδικασίες εγκληματικής κατηγορίας καθώς επίσης και συγκεκριμένες προϋποθέσεις έτσι όπως αυτές αναφέρονται στα γράμματα α και β του άρθρου 5. Στην κατάσταση αυτή φαίνεται ότι ε, ε, και βάσει και των ε, αποφάσεων της, του Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δεν μπορεί να υπάρξει νομιμοποίηση ε, ε, μπορεί ε, να καλυφθούν από μερικές όμως περιπτώσεις σύμφωνα και με την υπόθεση Butler όπου όμως δεν υπάρχουν ποινικέ καταδίκες. Στην περίπτωση Butler δεν έχουμε καμία ε, ποινική, ε, κανένα ποινικό αδίκημα το οποίο να αφορά οποιονδήποτε εμπλεκόμενο. Επίσης, ε, σε περίπτωση παρόμοια με την υπόθεση Butler, όπου δεν έχουμε ποινικό αδίκημα, μπορεί να θεωρηθεί ότι δεν μπορεί να εφαρμοστεί, και αυτό είναι το ερώτημα του Κοινοβουλίου που μου έχει υποβληθεί, να μην, θεωρηθεί το ε, το τεκμήριο της ε, ε, αθωότητας στην προκείμενη περίπτωση αυτό προϋποθέτει ότι υπάρχει ποινική υπόνοια κατά του ενδιαφερομένου. Και αυτό αντιτίθεται βεβαίως στο άρθρο 6 παράγραφος 2 ε, του, της ε, ε, Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων όσον αφορά τώρα την επαναχρήση των, δημευθέντων ε, ε, περιουσιακών στοιχείων. Σε μερικές περιπτώσεις και σε μερικές χώρες υπάρχουν διατάξεις οι οποίες αφορούν την επανάχρηση για ε, λόγους κοινωνικούς των προϊόντων δέσμευσης και δίμευσης προϊόντων εγκλήματος. Σε αυτήν την περίπτωση το εκτελών κράτος μέλος είναι αυτό το οποίο έχει την δυνατότητα να επαναχρησιμοποιήσει ε, τα ε, περιουσιακά αυτά στοιχεία. Θα πρέπει πάντως να υπενθυμίσουμε ότι τα όρια της, ε, των αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης καλύπτονται από τα όσα αναφέρονται στο 4 παράγραφος 1 της Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εν πάση περιπτώσει μονάχα μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων που παρέχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση βάσει του κανονισμού, βάσει της συνθήκης λειτουργίας μπορεί ε, να λειτουργήσει. Η παρούσα νομική βάση για την προτινόμενη οδηγία είναι τα άρθρα 82.2 και 83.1. Το άρθρο 82 παράγραφος 2 προβλέπει την έγκριση οδηγιών οι οποίες καθορίζουν κατελάχιστον ε, κανόνες όσον αφορά το αποδεκτόν των ε, ε, μαρτυριών και των αποδεικτικών στοιχείων, τα δικαιώματα των ατόμων όσον αφορά τις ποινικέ διαδικασίες και επομένως η χρήση των δεσμευθέντων και δημευθέντων προϊόντων δεν είναι δυνατόν να καλυφθούν από το άρθρο 82 ε, Το άρθρο 83.1 αναφέρεται στην έγκριση των οδηγιών οι οποίες καθορίζουν de minimis κανόνες όσον αφορά τον καθορισμό των ποινικών αδικημάτων καθώς επίσης ε, και των ε, ε, δυνατοτήτων άσκησης κυρώσεων. Όμως η επανάχρηση των δημευθέντων ή δεσμευθέντων περιουσιακών στοιχείων δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 83.1. Επομένως, το θέμα της επανάχρησης ε, των ε, δεσμευθέντων και δημευθέντων προϊόντων ε, εγκλήματος έτσι όπως αναφέρονται δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των άρθρων 82.2 και 83.1 του Κανονισμού Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης αν δεν συνάδουν δε ούτε με τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας. Επομένως, η απάντηση στο τέταρτο ερώτημα είναι ότι τα άρθρα 82.2 και 83.1 του Κανονισμού Λειτουργίας δεν ε, αποτελούν βάση για την ε, συμπερίληψη κανόνων και μέτρων όσον αφορά την επανάχρηση δεσμευθέντων και δημευθέντων ποσών και περιουσιακών στοιχείων. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα θα ήθελα να ζητήσω από όσους θέλουν να λάβουν το λόγο να είναι παρακαλώ όσο το δυνατόν συντομότεροι. Γιατί διαφορετικά ούτε στις 10 το βράδυ θα τελειώσουμε Όλοι θέλουμε να γυρίσουμε σπίτι νωρί, αλλά θέλουμε επίσης και να έχουμε αρκετό χρόνο για συζήτηση. Πραγματικά λοιπόν σας ζητώ να είστε σύντομοι. Εγώ έχω μια πολύ σύντομη ερώτηση για σας κύριε Καϊόλα. Είναι, με ναι ή όχι, απαντήστε παρακαλώ. Έχετε δει την τελευταία εκδοχή των συμβαστικών τροπολογιών που νομίζω της ε, συνταξαμε σήμερα αργά το πρωί ή νωρίς το μεσημέρι. Θεωρείτε ότι το κείμενο των συμβιβαστικών τροπολογιών εναρμονίζεται με τη νομική βάση. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Λάβαμε τις συμβιβαστικέ τροπολογίες μετά τις 12.30 το μεσημέρι και εκ πρώτης όψεως, έτσι πολύ σύντομα, βρίσκουμε δύο προβλήματα, δύο κύρια προβλήματα. Το ένα δεν έχει να κάνει με την νομική βάση, αλλά με τη χρήση του όρου σύσταση, recommendation. Σε αυτές τις διατάξεις μας φαίνεται ότι αυτός ο όρος δεν συνάδει με ένα καλό νομοθετικό κείμενο Το άλλο πρόβλημα, πιο σοβαρό, που εντόπισα είναι η συμβαστική τροπολογία 9. Εκ πρώτη όψεω, βέβαια, θα σα μιλήσω. Ε, τόσο αν θέλετε να επανέλθω και να το εξετάσω. Όχι, μάλιστα. Παρακαλώ να μας απαντήσετε τώρα. Ευχαριστώ πολύ. Μάλιστα, εντοπίσετε λοιπόν το πρόβλημα στα κριτήρια τα οποία βασίζονται στην ομολογία του Δικαστηρίου των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Θα ήθελα να, να τονίσω ότι τα κριτήρια Engel σκοπεύουν να απαντήσουν στην ερώτηση των ελάχιστων εγγύσεων σε περίπτωση ποινικών ε, διαδικασιών βασισμένα στο άρθρο, ε, σε περίπτωση που εφαρμόζεται το άρθρο 6 δεν εμπίπτει στα άρθρα 82 και 83 των συνθήκων. Στην υπόθεση Έγγελ ήταν μια πειθαρχική καθαρά προσφυγή. Άρα το δικαστήριο έπρεπε να λάβει υπόψη αυτή την πειθαρχική διαδικασία ε, σαν να επρόκειτο για ποινικό. Άρα δεν μπορούμε να μεταφέρουμε κάτι το οποίο δεν είναι ποινικό και να το μετατρέψουμε σε ποινικό. Αν δεν κάνω λάθο όμως, υπάρχει ένα άρθρο 3 στη τροπολογία συμβιβασμού που υποτίθεται ότι αντιμετωπίζει αυτό το θέμα. Η παράγραφος αυτή από τη δική μας άποψη δεν είναι καθόλου σαφής για να είμαι ειλικρινής. Την έχω εδώ μπροστά μου και δεν κατανοούμε τι σημαίνει και τι προαπαιτεί. Γιατί για παράδειγμα σημαίνει ότι τα κράτη-μέλη τα οποία προβλέπουν από το αστικό δίκαιο ότι η διαδικασία κατάσχεσης μπορεί να την εφαρμόσουν αν το επιθυμούν. Δεν είναι σαφές από τη διατύπωση. Πρόεδρος, εντάξει, εντάξει χρειάζεται χρήση διασάφησης. Πρόεδρος. Η κυρία Μακοβέη, η συγγήτρια. Ευχαριστώ. Το πρώτο τμήμα είναι απαρχαιωμένο, διότι αφορά ζητήματα τα οποία δεν υπάρχουν πλέον στην έκθεση και ιδιαίτερα ως προς την ισορροπία πιθανοτήτων τη στάθμιση πιθανοτήτων, γιατί μιλάμε για δίμευση όταν έχουμε να κάνουμε με μία ποινική καταδίκη και επιπροσθέτως μπορείτε να δημεύσετε περισσότερα με βάση το, το συγκεκριμένο αδίκημα και ανάλογα από τα στοιχεία ενεργητικού του προσώπου. Αυτό ισχύει από το 2005, από, συμβολή, από την απόφαση Συμβουλίου. Άρα αυτοί, αυτές οι δημεύσεις ε, διέπονται από τη στάθμιση πιθανοτήτων. Στην ε, τροπολογία Συμβασμού 9 που καλύπτει το άρθρο 5, δηλαδή πριν από την καταδίκη, δίμευση πριν από την καταδίκη αναφερόμαστε στη δίκαιη δίκη όπως ορίζει και το Συμβούλιο της Ευρώπης και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων όπως ισχύει σε κάθε περίπτωση ποινικού δηλαδή ο εναγόμενος να μπορεί να προσαχθεί δίκαια ενώπιον της δικαιοσύνης και αυτό ε, με βάση και την, ε, το χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων. Άρα δεν έχω και πολλά να σχολιάσω. Νομίζω ότι δεν δίδεται μία απάντηση, αλλά δεν θα ήθελα να μπω σε λεπτομέρειες. Θα ήθελα να πω ότι αυτό το, αυτά τα κριτήρια Engel δεν αναφέρονται ως κριτήρια απόφαση στην υπόθεση Engel. Δηλαδή, τα κριτήρια αυτά ενυπάρχουν στο κείμενο, μεταξύ άλλων. Μεταξύ άλλων. Και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για πολλά χρόνια λέει ότι εάν μία χώρα υπάγεται σε αυτό το καθεστώς πειθαρχικής δίωξης θα πρέπει να δούμε κατά πόσο είναι ποινική η υφής. Δηλαδή αν υπάρχουν εχέγγυα για να εναχθεί με βάση το ποινικό. Δηλαδή πρέπει να προχωρήσουμε πέραν από αυτά που ε, ορίζει και που ε, ζητά η νομική υπηρεσία. Παράγραφος 3 ε, τροπολογία συμβασμού 9 σημαίνει ότι οι χώρες που χρησιμοποιούν ένα διαφορετικό σύστημα μπορούν να το κρατήσουν. Για την κοινωνική επαναχρησιμοποίηση και για τη σύσταση στο άρθρο 1 παράγραφος 1 Μιλάμε για γενικές αρχές για την διαχείριση ε, των δημευθέντων ε, περιουσιακών στοιχείων και θα ήθελα η Σόνια να μιλήσει επί του θέματος διότι είναι ο τομέας της και βασίζεται και στην τροπολογία Μπορσαλίνο. Ένας ζητά το λόγο, δύο από τους σοσιαλιστές κάποιος. Ήσασταν ε, πολύ σύντομοι και σαφείς. Αλλά οι νομικές ε, διαφορές δεν έχουν επιληθεί. Η κυρία Αλφάνο καταρχήν. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ την Μόνικα για αυτή την ε, εξαιρετική εισήγηση σε σχέση με την επαναχρησιμοποίηση για κοινωνικούς σκοπούς των δημευθέντων στοιχείων ενεργητικών, δεν ξέρω κατά πόσο η νομική υπηρεσία μπορεί να χαλάσει αυτή την ισορροπία κατά τόσο έντονο τρόπο. Θα πρέπει λοιπόν να βάλουμε μια νέα αιτιολογική σκέψη για την ε, επαναχρησιμοποίηση υπό την ευρεία έννοια θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι πρόκειται για κάτι το αποτελεσματικό ε, ως προς την δίμευση στοιχείων ενεργητικού. Εφόσον δεν πρόκειται για δεσμευτικές διατάξεις, νομίζω ότι μπορούμε να δώσουμε το πολιτικό μας στίγμα δηλαδή την, τον πολιτικό μας προσανατολισμό που να οριοθετεί καλύτερα το ζήτημα ε, κατά τρόπο εμβληματικό. Και επειδή έχουμε εκφραστεί κατά αυτό τον τρόπο ως Κοινοβούλιο υπέρ αυτής της πρακτικής με βάση την ε, πλατφόρμα ΑΡΟ Μέσω αυτής της πλατφόρμας καταρτίζουμε βέλτιστες πρακτικές. Τη στιγμή που ο Συμβασμός ζητά από τα κράτη-μέλη να εγκρίνουν τα κατάλληλα μέτρα με βάση την προϋπάρχουσα πείρα για την ε, νέα χρήση δημευθέντων στοιχείων ενεργητικού, για σχέδια και προγράμματα πρόληψης του εγκλήματος, καθώς και έργα δημόσιας, δημόσιας ωφελίας και κοινωνικής ωφελίας, και εφόσον ζητάμε από τα κράτη-μέλη να μην δεχτούν εγκληματικά στοιχεία σε αυτή τη φάση, θα πρέπει να αποστείλουμε ένα πολιτικό μήνυμα για να μελετήσουμε μία νομική βάση έτσι ώστε στο μέλλον να είμαστε ακόμα πιο σαφείς και πιο αποτελεσματικοί. De Jong. Ευχαριστώ. Δύο ή τρία θέματα θα ήθελα να θίξω και εγώ. Τροπολογία Συμβασμού 7 που άλλαξε εκ νέου. νωρίς σήμερα το απόγευμα και που δείχνει και που αναφέρει ότι μετά μία απόφαση Εθνικού Δικαστηρίου, μετά από από ε, διαδικασίες, μετά από την διαδικασία, θα πρέπει να δούμε κατά πόσο η συγγήτρια θα ήθελε να δώσει μια καλύτερη μορφή ε, σε σχέση με την διαδικασία απόφασης, δικαστικής απόφασης. Αυτό θα μας βοηθούσε ιδιαίτερα. Μετά αυτά που είπε η νομική υπηρεσία για το 9, αυτή είναι η ουσία του ζητήματος. Συμφωνώ με τη Μονίκα Μακοβέη ότι δεν υπάρχουν πια, δεν υπάρχει στάθμιση των πιθανοτήτων. Και αφού διάβασα τη γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας, πιστεύω ότι αν και ισχύει ότι ε, ε, θα πρέπει να δούμε κατά πόσο έμεσα το άρθρο 6 ισχύει, θα πρέπει να δούμε κατά πόσο πρόκειται για ε, ποινικό, για καθαρά ποινικό δίκαιο ή όχι. Η διατύπωση λοιπόν θα μπορούσε να είναι καλή μέχρι του παρόντος και να δούμε σε ένα τριμερή διάλογο κατά πόσο πρέπει να επανασυντάξουμε. Προς το παρόν όμως χαίρομαι για το πώς, έχουν, πώς έχει το ζήτημα και η, ως προς την παράγραφο 3 ε, εγώ θα την διατύπωνα κάπως διαφορετικά. Δηλαδή τα κράτη-μέλη ε, διαθέτουν την επιλογή ε, συγκεκριμένων δράσεων και μέτρων ποινικού δικαίου. Και τέλος, συμφωνώ με την νομική υπηρεσία όταν πρόκειται για την επαναχρησιμοποίηση στοιχείων ενεργητικού και κερδών από συγκεκριμένες δραστηριότητες, διότι ζητάμε από τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν μία νομοθεσία. Δεν πρόκειται για ένα ψήφισμα ε, όπου αναφέρουμε ό,τι θέλουμε τι μας αρέσει και τι δεν μας αρέσει από τα κράτη-μέλη. Υπό αυτή την έννοια νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε κατά πόσο θα πρέπει να τεθεί κάτι τέτοιο στο ε, προήμιο. Δεν ξέρω λοιπόν κατά πόσο θα πρέπει να ενταχθεί στο λειτουργικό σκέλος της οδηγίας. Είμαι πολύ εντυπωσιασμένος από την εργασία που επετεύχθη και θα ζητήσω από την ομάδα μου να εγκρίνει. Η κυρία Σαρτζεντίνη. Ευχαριστώ. Θα είμαι ιδιαίτερα σύντομη και θα σταθώ μόνο στο εξής. Δηλαδή μπορούμε να μετατρέψουμε το αστικό δίκαιο σε ποινικό. Οι πράσινοι πιστεύουν ότι δεν θα πρέπει να δώσουμε ένα νέο ορισμό. Έχουμε πολλές αμφιβολίες για το κατά πόσο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το αστικό δίκαιο ως ποινικό. Ο κύριος De είπε ότι αυτός είναι ένας τρόπος προς τα εμπρός. Στο τριμερή διάλογο θα δούμε κατά πόσο μπορούν να επέλθουν αλλαγές. Αλλά αυτό είναι ανησυχητικό Κατέμε. Νομίζω ότι θα έχουμε εντολή να μπούμε σε τριμερή, αλλά αυτός ο τριμερής διάλογος θα είναι πολύ ασταθής. Και ε, τη στιγμή που θα είμαστε ασταθείς δεν θα μπορούμε και να ανταποκριθούμε. Δεν ξέρω κατά πόσο θα πρέπει να πιστέψουμε στο Συμβούλιο. Το εμπιστευόμαστε, ναι ή όχι. Το γεγονός ότι δεν λάβαμε υπόψη τα, τις δηλώσεις της δικής μας νομικής υπηρεσίας και έχουμε δύο διαφορετικά ε, γνωμοδοτικά κείμενα δικαίου δημιουργεί πρόβλημα. Η κυρία Μακουβέη. Ευχαριστώ, θα είμαι πολύ σύντομη Θα ήθελα να πω ότι δεν υπάρχουν διαφορές μεταξύ της νομικής υπηρεσίας και των τροπολογιών όπως διαμορφώνονται σήμερα. Ως προς το άρθρο 6 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και της Χάρτας θεωρούμε ότι θα πρέπει να δούμε ποια είναι η διατύπωση που χρησιμοποιείται στο ποινικό σε σχέση με τη δίμευση πριν από την καταδίκη. Και με βάση αυτά που είπε ο κύριος Ντεγιόγκ, θα προσθέσω αυτά τα στοιχεία, αλλά αν πρόκειται για δίμευση της περιουσιακής, ε, της περιουσίας, δεν σημαίνει ότι δεν θα υπάρχει και μια σχετική απόφαση, δικαστική απόφαση. Θα σας διαβάσω το κείμενο μετά από την δίκη σε σχέση με, μια ποινική, με ένα ποινικό έγκλημα θα πρέπει να γίνεται δίμευση με βάση απόφαση, δικαστική απόφαση. Και νομίζω ότι έτσι όλοι είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι. Ελπίζω πάντα να ήμασταν εξίσου ικανοποιημένοι με όλα τα θέματα, λέει η Πρόεδρος. Θα προσπαθήσω να συνοψίσω την κατάσταση και ξαναβάζω στη συζήτηση την πρόταση που έγινε προηγούμενα σήμερα το απόγευμα την κυρία Αλφάνο ε, να λάβει χώρα η ψηφοφορία για το θέμα της κυρίας Μακοβέη αύριο στις 9 και όχι στις 3. Δεν ξέρω τι σκέφτεται η συγγήτρια, πάντως να πω ότι διαπιστώνω ότι ακόμα και μετά τη συζήτηση η Νομική Επιτροπή δεν είναι ικανοποιημένη με τις συμβαστικές τροπολογίες. Ε, διαπιστώνω, διαβλέπω αυξανόμενη συνένεση μεταξύ των πολιτικών ομάδων, άρα εάν συνεχίσει η προσπάθεια ε, ίσως να φτάσουμε σε καλύτερο συντονισμό. Τέλος, όσον αφορά την ψηφοφορία, να σας πω ότι είδαμε πρώτα την ημερήσια διάταξη. Δεν είναι τόσο εύκολο, γιατί η ψηφοφορία αυτή ε, μαζί με άλλες δύο ε, προβλέπεται να κρατήσουν 17 ε, λεπτά. Επίσης υπάρχει και άλλο ένα στοιχείο ότι ζητήσαμε από την, ε, την κυρία Φλασίκοβα ε, Μπενόβα, η οποία είναι η συγγήτρια της συνέχεια που έχει στην εκχώρηση, στην εκχώρηση μαθητικών αρμοδιοτήτων κλπ. κλπ που είχε υποβληθεί ε, που είχε προγραμματιστεί για τις 9, εάν μπορεί να κάνει την παρουσίασή της στις 9.30 ή μάλιστα και το απόγευμα έτσι ώστε να έχουμε περισσότερο χρόνο. Ακόμα περιμένουμε την απάντησή της. Τέλος, το ΕΛΚ ζήτησε να προχωρήσουμε σε ψηφοφορία. Η εισηγήτρια όμως θα μας πει. Συμφωνείτε καταρχήν ε, να λάβει χώρα η ψηφοφορία από τις εκθέσεις αύριο στις 9.30 και όχι στις 3 το απόγευμα. Uh, Μπερδεύτηκα λίγο, λέει η κυρία, λέει η συγγήτρια κυρία Μακοβέη. Also that many people maybe they... ε, ναι, αλλά είπατε ότι και στις 9 ίσως α, ε, θα έρθουν, αλλά δεν θα ξέρουν ότι θα λάβει χώρα η ψηφοφορία. Ε, ε, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να είμαστε όσο γίνεται περισσότεροι, όσο περισσότεροι βουλευτές να είναι παρόντες. Και εγώ το νομίζω, λέει ο Πρόεδρος. Αλλά εδώ έχω ένα χαρτί Έχω ένα χαρτί λοιπόν που λέει ότι αύριο στις 9 θα έχουμε πρώτα την έκθεση της κυρίας Φλασίκοβα Βαμπένοβα και μετά στις 9.30 έχουμε την παρουσίαση του τρίτου κοινού υποπτικού οργάνου της Ευρωπόλ, τη FTP και μετά έχουμε και κάτι άλλο. Δεν προβλέπεται ψηφοφορία για τις 9 το πρωί. Α, λέτε ότι η ψηφοφορία θα γίνει στην κρίμα αύριο. Α, τότε μπερδεύεται ακόμα περισσότερο. Δεν έχω τίποτα, ε, καμία σχέση με την κρίμα, αλλά ζήτησε η πρόεδρος της ε, Κρίμε να λάβει χώρα η, Λίμπε, ε, η ψηφοφορία στη Λίμπε 9 το πρωί. Η κυρία Αλφάνο, η πρόεδρος της Κρίμε, ίσως μπορεί να μας πει σε 30 δευτερόλεπτα τι εννοεί. Λοιπόν, λαμβάνοντα υπόψη ότι η Μόνικα είναι εδώ, να σας, να, σας εξηγήσω και να τις εξηγήσω. Λοιπόν, αύριο το απόγευμα στις 3 προβλέπονται οι ψηφοφορίες στη ΛΥΜΠΕ. Όμως, ταυτόχρονα, στην Επιτροπή ΚΡΙΜ έχουμε μία δραστηριότητα που έλεγε, όπως έλεγε και η Στάνφος Βερονίκ, μας έχει απασχολήσει τους τελευταίους μήνες, μετά από ε, ε, πρόσκληση που απίθυνε ο πρόεδρος Σούλτσε σε εκπροσώπους άλλων κοινοβουλίων, καθώς επίσης και στην επίστροπο Μάλστρομ. Πρόεδρος, δεν με ενδιαφέρει τι θα κάνετε στην Κρίμ. Εσείς προτείνετε ναι ή όχι να λάβει χώρα ψηφοφορία αύριο 9 το πρωί. Ε, και θέλετε να μας πει την άποψή της εισηγήτρια ναι ή όχι. Μα αυτό είπα όταν ξεκίνησε η συνεδρίαση. Ζήτησα λοιπόν ε, στις 3 η ώρα ήδη, εάν είναι δυνατόν, αντί να λάβει χώρα η ψηφοφορία αύριο στις 3, ε, ε, στις 9 το πρωί ή στις 10.30-11 το πρωί. Παρότι είπα, ήδη στην Επιτροπή Κρίμα έχουμε προβλέψει κάποιες ε, κάποιες ε, ε, άλλες ψηφοφορίες. Λοιπόν, 9 το πρωί θα, αν, αν συμφωνείτε να γίνει ψηφοφορία στη Λίμπε. Σορτζεντίνη. Ναι, γι' αυτό ακριβώς μου ζήτησαν και οι συνεργάτες μου να έρθουν εδώ. Λιγότερο από 24 ώρες λιγότερο από 24 ώρες πριν από την ε, ψηφοφορία. Ε, δεν μπορούμε να είμαστε σε δύο μέρη ταυτόχρονα και τι να σας πω τώρα, πιστεύουμε ότι τέτοιου είδους αιτήματα θα πρέπει να προωθούνται ε, μέσω των συντονιστών. Ζητώ λοιπόν να μην υποκύπτουμε σε τέτοιου είδους ε, ε, αιτήματα, γιατί κινδυνεύουμε να μην έχουμε όλους όσους επιθυμούμε παρόντες στην στιγμή της ψηφοφορίας. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να αλλάξει αυτή η κατάσταση. Η κυρία Ματιέ. Η κυρία Ματιέ θα πάρει το λόγο. Δεν μπορώ να σας ξαναδώσω κυρία Αλφάνο το λόγο. Μπερδευτήκαμε λίγο. Κοιτάξτε. Έχουμε αυτή την Επιτροπή κρίμα η οποία η οποία πρέπει έχει αναλάβει πάρα πολύ δουλειά να κάνει και πρέπει να τη βοηθήσουμε και λίγο. Έχουμε την ενδιάμεση έκθεση της ΚΡΙΜ, η οποία φτάνει στην ψηφοφορία. Ε, είχαμε 700 τροπολογίες ε, στην έκθεση. Ο εισηγητής ε, συζητάει αυτή τη στιγμή, οι συμβασικές τροπολογίες θα ψηφιστεί η έκθεση αυτή αύριο. Ωραία. Η Επιτροπή ΚΡΙΜ λέει ότι μπορεί να προσαρμόσει τις, ε, ε, το ωράριο ψηφοφορίας της ε, με την προϋπόθεση ότι και η ΛΥΜΠΕ θα κάνει μια μικρή προσπάθεια. Τώρα, αν θέλετε, ε, μπορούμε να συζητήσουμε και την Πέμπτη, αλλά την Πέμπτη είναι η ε, ανάληψη και ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι την Τετάρτη το απόγευμα πριν από την Πέμπτη της αναλήψεως κανείς δεν πρόκειται να έρθει να ψηφίσει ούτε στη Λίμπε ούτε στην Κρίμ. Και επομένως πρέπει να ξέρουμε ότι την Τετάρτη απόγευμα δεν παίζει καμία ψηφοφορία. Εάν θέλουμε πραγματικά να έχουμε, ε, ε, να έχουμε ψηφοφορίες, θα πρέπει οπωσδήποτε να λάβουν χώρα και οι δύο ψηφοφορίες το πρωί της Τετάρτης. Μα δεν μιλάμε για την Τετάρτη, μιλάμε για την Τρίτη. Ναι, αλλά ξέρετε ότι ε, σε πολλές χώρες ε, και η Τετάρτη είναι αργία. Εάν θέλουμε, εάν θέλουμε παρουσία βουλευτών, ε, θα πρέπει να έρθει να γίνουν οι ψηφοφορίες την Τρίτη. Τη Δευτέρα είναι όλοι εδώ. Ε, την Τρίτη επίσης είναι πάρα πολύ εύκολο να ζητήσουμε τους βουλευτές να είναι παρόντες και να κάνουν δύο ψηφοφορίες, μία στη Λίμπη και μία στην Κρίμ. Δεν είναι και τίποτα τρομερές ε, ψηφοφορίες και νομίζω ότι με τον τρόπο αυτό και θα βοηθήσουμε τις επιτροπές και θα μπορέσουμε να ε, προωθήσουμε τα θέματά μας. Η κυρία Μακοβέη. Ευχαριστώ. Η κυρία Αλφάνο έκανε μια πρόταση με ρωτάτε εάν με ρώτησε. Ναι, με είχε ρωτήσει και εγώ συμφωνώ. Και λαμβάνοντας ε, υπόψη την ευελιξία της ΚΡΙΜ και μια και είμαι και εγώ η ίδια ε, ε, μέλος της ΚΡΙΜ, προτείνω να ξεκινήσουμε εδώ με την, με την ε, ΛΥΜΠΕ. Ναι, δεν, δεν είπα εγώ τι ώρα. Είπαμε, είπα να ψηφίσουμε πρώτα στην ΛΥΜΠΕ, άρα στις 9 και μετά στην ΚΡΙΜ. Ναι, αλλά αυτό σημαίνει ότι ε, γίνεται μεγάλο μπέρδεμα λέει η Πρόεδρος. Δεν συζητάμε να ψηφίσουμε την Τετάρτη. Λέει η κυρία Αλφάνο ότι αντί να ψηφίσουμε στις 3 το απόγευμα να ψηφίσουμε το πρωί της Τρίτης. Εγώ δεν είμαι καθόλου ευτυχής ε, να ε, συζητάμε τέτοια πράγματα εκτός των συντονιστών. Δεν μου αρέσει καθόλου που υπάρχουν τα αιτήματα αυτά για αλλαγές. Θέλω να το δουν οι συντονιστές. Εγώ δεν πιστεύω ότι πρέπει να αλλάξει η ψηφοφορία Καταλαβαίνω ότι η κυρία Μακοβέη είναι, ε, είναι διαθέσιμη. Ναι, αλλά μας λένε, λέει η κυρία Μακοβέη, ότι τρεις η ώρα θα έρθει η Επίτροπος Μάλστρομ και ένα σωρό βουλευτές ε, από τα Εθνικά Κοινοβούλια. Ναι, αλλά λέει η Πρόεδρος, εμείς έχουμε καθορίσει την ψηφοφορία μας αύριο, αύριο Τρίτη, όχι μεθαύριο Τετάρτη, αύριο Τρίτη στις 3. Και ούτε σε άλλους δεν θέλω να συζητάμε και ε, διαρκώς για το θέμα αυτό, γιατί όλοι έχουμε και κάποια άλλη δουλειά. Κοιτάξτε, ε, έπρεπε να είχε συζητηθεί το θέμα και να είχε ολοκληρωθεί πριν. Ε, ε, εγώ νομίζω ότι πρέπει να σταματήσει η συζήτηση. Ε, θα πρέπει οι συντονιστές να αποφασίσουν με συνεννοούμενοι μέσω ηλεκτρονικού ταχυδραμείου. Εάν οι συντονιστές πιστεύουν ότι θα πρέπει αύριο στις 9 να λάβει χώρα ψηφοφορία στη ΛΥΜΠΕ ε, και ότι όλα τα άλλα σημεία της ημερήσιας διάταξης μπορούν να ε, συζητηθούν σε άλλες ώρες, γιατί και αυτό δεν είναι δεδομένο, τότε, τότε εντάξει να γίνει η ψηφοφορία αύριο 9 η ώρα το πρωί. Δεν μπορούμε τελικά ε, λίγο πριν την παρουσίαση τη εκθεσή του, να πούμε στου συζητητές «Α, όχι, ξέρετε, δεν μπορείτε τώρα να, μην, να συζητήσετε την έκθεσή σα. Ε, λοιπόν, νομίζω ότι δεν υπάρχει λόγο να συνεχίσουμε τη συζήτηση. Κυρία Ματιό, δεν καταλαβαίνω γιατί θέλετε ξανά το λόγο. Γιατί δεν μπορούμε να ψηφίσουμε, λέει η κυρία Ματιό. τι, να συνεδριάσουν οι συντονιστές. Άμα δεν υπάρχει συνεδρία συντονιστών, εσύ δεν είπατε, εσείς δεν το είπατε. Κυρία Ματιό, κυρία Ματιό, έχει τελειώσει, έχει λήξει το θέμα. Με συγχωρείτε λοιπόν γι' αυτό. Για τη σύγχυση που δημιουργήθηκε θα προχωρήσουμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Συγγνώμη, δεν κατάλαβα τι είπατε, κυρία Αλφάνο. Πρόεδρος, ναι, νομίζω πως αυτό πρέπει να διευθετηθεί από τους συντονιστές των πολιτικών ομάδων. Αυτό είναι και το έργο τους εξάλλου διότι... Δεν είναι Κοιτάξτε, δεν είναι δημοκρατική αυτή η διαδικασία, ε, λέει η κυρία Αλφάνο. Όχι, όχι, αυτή είναι η διαδικασία. Δεν είναι, δεν είναι σωστό αυτό που λέτε, ούτε αυτό που λέει η συνάδελφος είναι σωστό. Όχι, το θέμα έληξε, λέει η πρόεδρος. Προχωρούμε λοιπόν στα προσωπικά δεδομένα. Εισηγητής ο κύριος Άλμπρεχτ, ο οποίος δεν είναι εδώ. Μάλιστα, διακοπή 10 λεπτών τώρα. Θα μπορέσουμε λοιπόν να συζητήσουμε οι συντονιστές. Αρχίζουμε 5 παρατέταρτο με την έκθεση για τα προσωπικά δεδομένα του κυρίου Άλμπρεχτ. Okay, Συνάδελφοι, συνεχίζουμε. Καταρχάς, να σας πληροφορήσω ότι η μερίσια διάταξη θα παραμείνει ως έχει. Παρακαλώ καθίστε. Η μερίσια διάταξη παραμένει ως έχει. Τώρα, προχωρούμε λοιπόν στον κύριο Άλμπρεχτ, ο οποίος κουβεντιάζει βλέπω. Κύριε Άλμπρεχτ, είστε έτοιμος. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς, θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη, διότι αυτή η αναβολή έτσι οδήγησε σε κάποιες ε, απουσίες των ε, σκιωδών εισηγητών, κάποιων από αυτούς που δεν μπορούσαν να είναι εδώ σήμερα. Ελπίζω όμως να μην δημιουργήσει αυτό σημαντικά προβλήματα για ορισμένε κοινοβουλευτικέ ομάδες σήμερα σε αυτήν την συνεδρίαση. Όταν προγραμματίσαμε τη συνεδρίαση αυτή, ε, σκεφτήκαμε πως θα έπρεπε να έχουμε μια άλλη ανταλλαγή απόψεων εδώ στην Επιτροπή για τις τροπολογίες και τα διάφορα σημεία που θίγησαν, διότι υπάρχουν τόσες πολλές τροπολογίες, τόσα πολλά ζητήματα τα οποία πρέπει να επιληθούν, που πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να συζητηθούν ξεχωριστά. Την τελευταία φορά δεν μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό επειδή πάλι έλειπαν αρκετοί. Και τώρα πάλι ο κύριος Φως, η κυρία Πλάτφορντ και οι υπόλοιποι σκιώδεις οι και ο κύριος Δρούτσας από τους σοσιαλιστές δεν μπορούν να έρθουν σήμερα και αυτό με οδηγεί στο να πω ότι σήμερα μπορώ μόνο να απαντήσω σε ερωτήσεις και να ακούσω τους προβληματισμούς σας και να τους μεταφέρω λοιπόν, καθώς και αυτήν την ανταλλαγή απόψεων στους σκιώδεις εισηγητές, διότι θα συναντηθούμε αύριο. Θα, και να σας ενημερώσω τώρα λοιπόν για το πού βρισκόμαστε. Ε, έγιναν 4 ή πέντε συνεδριάσεις των σχεδόν εξηγητών μέχρι τώρα. Όπως σας είπα, τροπολογίες είναι πάρα πολλές, τα άλλα τα θέματα είναι πάρα πολλά. Δεν καταφέραμε να κάνουμε τις ε, συνομιλίες που θέλαμε να κάνουμε, όσες θέλαμε. Χρειαζόμαστε λίγο χρόνο ακόμα επομένως και πιστεύω ότι δεν θα καταφέρουμε να ψηφίσουμε στις 29 Μαΐου, καθώς φαίνεται, με αυτούς τους ρυθμούς. Από πλευράς μας λοιπόν πρέπει να αναβάλουμε την ψηφοφορία σε εκείνη τη συνεδρίαση. Εξακολουθούμε φυσικά σαφέστατα να επιθυμούμε να ολοκληρώσουμε αυτούς τους δύο φακέλους, τον κανονισμό και την οδηγία την οποία θα συζητήσουμε αύριο. Και τα δύο πρέπει να ψηφιστούν μαζί πριν την διακοπή για καλοκαίρι. Προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε να δρομολογηθεί αυτό το συντομότερο δυνατόν. Θα χρειαστούμε όμως μερικές επιπλέον συναντήσεις. Αύριο θα συναντηθούμε για τις θυμιβαστικές ε, τροπολογίες. Πιστεύω πάντως σε γενικές γραμμές ότι κάνουμε τεράστια πρόοδο. Τελευταία συνάντηση ήταν πάρα πολύ καλή. Είχαμε αρκετές ε, ε, θέσεις τις οποίες καταλήξαμε, κατορθώσαμε να συμβιβαστούμε. Ήταν δύσκολο να καθορίσουμε μια ενιαία γραμμή. Όπως θα, δείτε τα άρθρα συνδέονται μεταξύ τους ε, και αναφέρονται εξίσου σε πολλούς τομείς, το πεδίο εφαρμογή τους, σε κανόνες σχετικά με τη συγκεκριμένη επεξεργασία δεδομένων και τη διαδικασία ε, που αυτό δεν μπορεί να, ε, να αναλυθεί ξεχωριστά από τα ατομικά δικαιώματα. Μετά το θέμα των υπαλλήλων που επεξεργάζονται τα δεδομένα σε γενικές γραμμές όμως να σας πω ότι θα ακολουθήσουμε τις γραμμές του ψηφίσματός μας ε, του Ιουλίου του 2011 όπου δώσαμε το στίγμα μας, είπαμε πού βρισκόμασταν, ακολουθήσαμε την ε, οδηγία του 1995 και είπαμε ότι δεν θέλουμε το σύστημα να αλλάξει ριζικά, δεν θέλουμε διαφορετικούς ε, κανόνες, αλλά αυτό που θέλουμε είναι σε γενικέ γραμμέ τα ίδια, αλλά μια ενιαία εναρμονισμένη νομοθεσία. Αυτή είναι η γραμμή μας, η κύρια γραμμή μας. Και επίσης θέλουμε να συνεισφέρουμε και να συμπεριλάβουμε την εμπειρία που έχουμε στον ε, τομέα της πληροφορικής τα τελευταία 10-15 χρόνια. Ελπίζω οι συμβιβασμοί να υιοθετηθούν με ευρεία ε, πλειοψηφία τον Μάιο. Όπως σας είπα όμως, θα συζητήσουμε και άλλο με τους σκιώδεις εισηγητές. Παρακαλώ εσάς να επικοινωνήσετε με τους κοιόδης εισηγητές σας και με εμένα να έχετε οποιαδήποτε ερώτηση ή προβληματισμό είτε κάποια σημεία που εσείς θέλετε να φέρετε στις ε, συζητήσεις μας. Εμπιστευτείτε τους κοιόδης εισηγητές σας, διότι αυτό που προσπαθούμε τώρα είναι να επιτύχουμε μία γενική συνένεση, έτσι ώστε να διευκολυνθεί και η ψηφοφορία σε όλες, όλες αυτές τις τροπολογίες. Δεν είναι εύκολο έργο, Πρέπει πραγματικά να προσπαθήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο να διευκολύνουμε το έργο αυτό τη ε, ψηφοφορία έτσι ώστε να οδηγηθούμε σε διαπραγματεύσει με το Συμβούλιο μέχρι το καλοκαίρι. Και πιστεύω ότι η Ιρλανδική Προεδρία κάνει μια εξαιρετική δουλειά. Προχωρούν καλά, με καλούς ρυθμούς και πιστεύω πως θα καταφέρουν να ψηφίσουν την διαπραγματευτική εντολή ή τουλάχιστον τη βάση της διαπραγματευτικής εντολής πριν διακόψουμε για καλοκαίρι ώστε να αρχίσουν οι διαπραγματεύσει αμέσως μετά τις καλοκαιρινές διακοπές. Σας ευχαριστώ πολύ για την... και χαίρομαι για την ανταλλαγή απόψεων. Ευχαριστώ πολύ κύριε Άλμπρεχτ. Ήδη μας ε, αναφέρατε ότι πολλά μέλη δυσκολεύτηκαν να παρευρεθούν σήμερα εδώ. Έχουμε λοιπόν πολύ λίγους κοιόδης εισηγητές εδώ. Νομίζω ο κύριος Βαντεκάμπ θα αντικαταστήσει τον κύριο Βόσα για το ΕΛΚ. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ιντφέλντ. Όπως, και, όπως είπε και ο Γιάνν Φίλιπ, ο Άξελ δεν μπορεί να, να είναι εδώ μαζί μας. Χαίρομαι που μπορώ να τον αντικαταστήσω και να τοποθετηθώ σε αυτήν την πολιτική συζήτηση. Η δική μου ομάδα ανέκαθεν τόνιζε ότι η προστασία δεδομένων είναι δικαίωμα των πολιτών και διευκολύνει την ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Αυτά συνάδουν. Και οι δύο πλευρές πρέπει να ενισχυθούν έτσι ώστε να έχουμε μια, προστασία, ε, μια νομοθεσία για την προστασία δεδομένων που να αντιμετωπίζει ε, που να έχει μεγάλο εύρος. Επίσης, για το ΕΛΚ ορισμένα σημεία είναι ιδιαίτερη σημασία. Καταρχάς, η μείωση της γραφειοκρατίας όσον αφορά την υποχρέωση κοινοποίηση και πληροφόρηση για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Έπειτα, να διευκρινιστούν οι ευθύνε και το, οι αρμοδιότητε των ε, ελεκτών και των, ε, και των όσων επεξεργάζονται τα ε, προσωπικά δεδομένα. Τρίτον, τα επιχειρηματικά μοντέλα. Τέσσερα, η χρήση των δεδομένων από τις ασφαλιστικές εταιρείες. Πέμπτον, η χρήση των δεδομένων για έρευνα. Έκτον, αυτορύθμιση για τις εταιρείες για μείωση της εγγραφειοκρατίας. Και τέλος, εις βάθος προτάσεις σχετικά με το δικαίωμα κάποιου να λησμονηθεί και το αν αυτό είναι τεχνικά εφικτό. Το ότι ζητάμε όλα αυτά δεν σημαίνει ότι τα δικαιώματα των πολιτών θα παραμεληθούν. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι η σωστή ισορροπία σε πολύ κέρια σημεία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Εκ μέρους των σοσιαλιστών, κυρία Ρωμέρο Λεόπες. Ε, Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ε, δεν μπορώ να μιλήσω ακριβώς εκ μέρους του Δημήτρη. Μου το ζήτησε βέβαια. Θα ήθελα όμως να χρησιμοποιήσω αυτό το βήμα για να θίξω ορισμένα σημεία. Και εγώ έχω υποβάλει προσωπικά κάποιες πρωτολογίες και θα ήθελα φυσικά να ε, τύχουν τις ε, συμφωνίες του εισηγητή. Η πρώτη είναι η τροπολογία 97 όπου αναφέρεται ότι κάποιος μπορεί να αποσύρεται στην κατάθεσή του για την χρήση των προσωπικών του δεδομένων Και τι γίνεται τώρα, όταν δίνει τη συγκατάθεσή σου, πολλέ φορέ είναι εύκολο να το κάνει. Είναι όμω πολύ δύσκολο να αποσύρει τη συγκατάθεσή σου. Τεχνικά μιλώντα. Πρέπει λοιπόν να διασφαλίσουμε αυτό να γίνεται απόλυτα κατανοητό και ο ενδιαφερόμενος να μπορεί να αποσύρει τη συγκατάθεσή του το ίδιο εύκολα με το να τη δώσει. Επίσης, μια άλλη τροπολογία που θα ήθελα να γίνει δεκτή από τον εισηγητή και τους συνεισηγητές είναι για τις εταιρείε που αποθηκεύουν αυτά τα δεδομένα, το τεράστιο ρυθμό δεδομένων, τις εταιρείε ε, του νέφους, τα cloud companies που λέμε. Πολλές φορές είναι υπεργολαβίες, λειτουργούν με τέτοιο τρόπο και φυσικά χρειάζεται η... το έργο αυτό να είναι από κάποιον που να έχει την ανάλογη ευθύνη Χρειάζονται λοιπόν και οι αντίστοιχες ρυθμιστικές διατάξει για την προστασία των δεδομένων και ως προς τις εταιρείες που τα διαχειρίζονται. Αυτό πρέπει να το φροντίσουμε πιστεύω έτσι ώστε να καλύψουμε την προστασία των δεδομένων από αυτές τις εταιρείε, από τις εταιρείε ενέφους. Επίσης, μια άλλη τροπολογία που για μένα είναι σημαντική είναι αυτή που αναφέρεται στην συνεκτικότητα όταν έχεις μια εποπτική ε, αρχή και μια εταιρεία η οποία είναι θηγατρική. Αυτό δημιουργεί προβλήματα. Για παράδειγμα, όταν, κάποιος, ένα, όταν ένα κράτος μέλος έχει πρόβλημα με μια εταιρεία η οποία λειτουργεί με θηγατρικές, η ελεκτική αρχή της κύρια ε, κύριας εταιρείας είναι αυτή που αναλαμβάνει την ευθύνη και αυτό πιστεύουμε πως είναι ένα προβληματικό σημείο, όχι μόνο ως προς την ερμηνεία του από τα διάφορα νομικά συστήματα. Η νομοθεσία, όπως ξέρετε, διαφέρει από κράτος μέλος σε κράτος μέλος. Αυτό που προτείνουμε είναι, εκτός από την ελεκτική αρχή στην ε, κύρια εταιρεία, να υπάρχει συντονισμός των δράσεων και των θεργατρικών. Αυτό λοιπόν το έργο του συντονισμού είναι πολύ σημαντικό και θα πρέπει να είναι αρκετό για την επίλυση τυχόν ε, προβλημάτων που προκύψουν. Χρειάζεται λοιπόν μια καλή ελεκτική αρχή από τα κράτη-μέλη του κράτους μέλους προέλευσης. Πιστεύουμε πως αυτό θα λύσει πολλά προβλήματα. Αυτό είναι μια πρόταση της Ισπανικής ε, Υπηρεσίας Προστασίας Δεδομένων, η οποία συνειδητοποίησε ότι ενδεχομένως υπάρξουν προβλήματα στο μέλλον και θα ήθελε λοιπόν αυτό να το λάβει υπόψη του ο εισηγητής και παρεμπιπτόντως να το συγχαρώ και για το εξαιρετικό του έργο και την συνέπεια με την οποία εργάζεται. Οι τροπολογίες είναι εξαιρετικές. Ευχαριστώ. Υπάρχουν άλλοι συνάδελφοι που θα ήθελαν να σχολιάσουν. Αν όχι, τότε θα πάρω εγώ το λόγο, πολύ σύντομα. Δύο σχόλια για το πεδίο εφαρμογή. Το πρώτο. Το πολύ λοιπόν, η πολύ συζητημένη προσέγγιση δέσμης. Δεν είμαστε σίγουροι. Ίσως μπορεί η Ιρλανδική Προεδρία να μας το διευκρινίσει, αλλά πιστεύουμε ότι τα κράτη-μέλη έχουν καταλήψει πλήρως την ε, ιδέα της ε, απόσυρση των δημόσιων υπηρεσιών από τον κανονισμό αυτό και να υπάγονται πλέον ε, στην κατηγορία, στην οδηγία, συγχωρείτε. Επίσης, όσον αφορά το πεδίο εφαρμογή, εμείς ανέκαθεν ζητούσαμε ένα, ένα ενιαίο μέσο. Γι' αυτό και η προσέγγιση δέσμης Πιστεύουμε λοιπόν πως οι δημόσιες υπηρεσίες πρέπει να συνεχίσουν να καλύπτονται από τον κανονισμό. Έπειτα, κάτι που πιστεύω πως είναι πάρα πολύ σημαντικό για όλα τα υπόλοιπα, ο ορισμός των προσωπικών δεδομένων. Ο ορισμός των προσωπικών δεδομένων θα είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ε, γίνεται πολλής λόγος για τα ανώνυμα δεδομένα, την ανωνυμοποίηση των δεδομένων. Εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχει τέτοιο πράγμα πλέον, διότι τα, όταν τα ανώνυμα δεδομένα συγκεντρωθούν, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να απομονώσουν συγκεκριμένα άτομα. Και δεν υπάρχει καμία διαφορά ή ελάχιστη διαφορά ως προς τον ε, εντοπισμό ενός ε, ατόμου μέσω της χρήσης ανώνυμων δεδομένων. Πιστεύω πως χρειάζεται να τροποποιήσουμε λοιπόν τις προτάσεις μας σύμφωνα με τα νέα δεδομένα που έχουμε και πραγματικά θα ήθελα να ακούσω του εμπειρογνώμονε να μας πούν, να μας ενημερώσουν. Δυστυχώ οι φόβοι μου επιβεβαιώθηκαν από τι απαντήσει του και πραγματικά πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό, να δούμε δηλαδή πώς χρησιμοποιούνται τα προσωπικά δεδομένα, πώς ορίζονται και αν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να απομονώσουν ένα συγκεκριμένο άτομο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό ως στοιχείο κλειδί για όλη την νομοθεσία που θέλουμε να περάσουμε. Τώρα θα ήθελα να ζητήσω από ε, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πάρει το λόγο αν το επιθυμεί, έπειτα από την Ιρλανδική Προεδρία και στο τέλος θα επανέλθουμε στον εισηγητή. Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ. Είμαι διευθυντή τη Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνη. είμαι υπεύθυνο για το θέμα αυτό. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία και να σας πω ότι εκτιμούμε πάρα πολύ το έργο που έχει γίνει από τους εισηγητέ εδώ στο Κοινοβούλιο. Είμαστε στη διάθεση των εισηγητών και στη διάθεση της ομάδας στο σύνολό της για οποιαδήποτε βοήθεια τεχνικής ή άλλης φύσης. Βλέπουμε κάποια στοιχεία προόδου παράλληλα στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο και είμαστε αισιόδοξοι ότι αυτές οι εξελίξεις θα καρποφορήσουν εν το χρόνο. Να σας πω ότι δεν θέλουμε να κάνουμε επανάσταση στην νομοθεσία, θέλουμε να την εξελίξουμε, γιατί πρόεδρος Ρέντινγκ έλεγε ανέκαθεν ότι πρώτον θέλουμε να βελτιώσουμε και την οδηγία και την απόφαση πλαίσιο ως προς την προστασία των, των πολιτών, αλλά και για την καλύτερη λειτουργία της ενιαίας αγοράς. Επίσης, η έκθεση ΒΟΣ του 2011 έτυχε ευρείας υποστήριξη στην Ολομέλεια και πραγματικά έδωσε το στίγμα του Κοινοβουλίου, τη θέση του Κοινοβουλίου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλωσόρισε αυτήν την νομοθετική πρόταση. Καλωσορίζουμε και το έργο όλων των ε, πολιτικών ομάδων, των ε, σκιωδών εισηγητών που βασίστηκαν στην έκθεση ΦΟΣ. Τώρα όσον αφορά το ισχύον καθεστώς προς το παρόν και τις δύο ερωτήσεις οι οποίες τέθηκαν από την Πρόεδρα. Θα ήθελα να πω, όσον αφορά αυτές, ότι φυσικά η συνθήκη στο άρθρο 72 αναφέρεται ρητά στον νόμο και την τάξη. Δεν θέλουμε να κάνουμε κάποια αλλαγή εκεί. Ταυτόχρονα όμως, η συνθήκη περιλαμβάνει και διάφορα άλλα κεφάλαια που αναφέρονται και στην οδηγία και στην απόφαση πλαίσιο όπου συμπεριλαμβάνονται σχεδόν τα πάντα εκτός από το ποινικό δίκαιο. Η απόφαση δηλαδή πλαίσιο αναφερόταν στο ποινικό δίκαιο και αυτό το βρίσκουμε λογικό. Και η δομή που έχουμε προτείνει τώρα, δηλαδή ένας κανονισμός για τα πάντα, εκτός από την οδηγία η οποία αναφέρεται στο κεφάλαιο που καλυπτόταν παλιότερα από την απόφαση πλαίσιο, είναι απολύτως εναρμονισμένη με την δομή της συνθήκης. Και φυσικά, το να μεταφέρουμε από τον κανονισμό στην οδηγία έναν ολόκληρο, ένα ολόκληρο κομμάτι του δικαίου είναι ασύλληπτο, διότι οι πολίτες θα μείνουν χωρίς καμία προστασία. Προστασία την οποία είχαν υπό την οδηγία που μέχρι τώρα ίσχυε. Δεν θεωρώ λοιπόν ότι μπορούμε να προχωρήσουμε τις συζητήσεις προς αυτό αυτή την κατεύθυνση. Αλλά πραγματικά αυτό που θέλω να τονίσω και να επαναλάβω είναι ότι το κύριο μέλημά μας είναι η προστασία των πολιτών και η καλύτερη προστασία των πολιτών και των ατομικών τους δικαιωμάτων, ιδιαίτερα σε μια εποχή που τα πάντα μπορούν να αποθηκευτούν, να συλλεχθούν και να διατηρηθούν εσάι μέσω του ίντερνετ. Όσον αφορά τώρα τα προσωπικά δεδομένα, ίσως θα έχετε δει ότι στην πρότασή μας έχουμε διατηρήσει τους κύριους ορισμούς της οδηγίας, αλλά είμαστε ανοιχτοί ε, σε διευκρινήσεις όσον αφορά τις ε, τεχνικές αναφορές, τα τεχνικά στοιχεία, ιδιαίτερα όσον αφορά τα ψευδόνυμα στοιχεία. Πιστεύουμε πως αυτά τα ψευδόνυμα στοιχεία πρέπει να καλύπτονται από τον κανονισμό και την οδηγία. Και πραγματικά, στις Ηνωμένε Πολιτείε έχουμε δει ότι τέσσερα στοιχεία, φύλλο, ηλικία, ταχυδρομικός κώδικας και κάτι άλλο που δεν θυμάμαι ακόμα, μπορούν να οδηγήσουν στον εντοπισμό και στην ταυτοποίηση 95% του πληθυσμού. Αυτά τα τέσσερα πράγματα λοιπόν. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να δούμε αν, μπορούμε, αν έχουμε το περιθώριο να κάνουμε εκπτώσεις λοιπόν όσον αφορά αυτά τα ψευδόνυμα δεδομένα. Από την άλλη όμως, όταν ένα άτομο μπορεί να εντοπιστεί, να απομονωθεί με τη χρήση αυτών των στοιχείων, τότε αυτό είναι κάτι που δεν καλύπτει ο κανονισμός και πρέπει πραγματικά να θέσουμε τα όρια. Να τραβήξουμε μία γραμμή. Αυτό θα ήθελα να απαντήσω στις δύο ερωτήσεις της Πρόεδρου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ρόρι Γκόγκαν εκ μέρους της Ιρλανδικής Προεδρίας τώρα έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Θα σας ενημερώσω σχετικά με το πού βρίσκεται το Συμβούλιο στη διαπραγματεύσεις αυτή την εποχή. Όπως γνωρίζετε, Είχαμε διεξάγει συζητήσει για τον κανονισμό για να μεγιστοποιήσουμε την πρόοδο που μπορούμε να επιτύχουμε. Έχουμε σχεδιάσει 20 συνεδριάσεις της DAPIX. Τις αυξήσαμε τώρα σε 26 ημέρες. Στις 6 Ιουνίου θα πάει το θέμα στο Συμβούλιο για να απαντηθούν ορισμένα βασικά ερωτήματα όσον αφορά αυτά τα τέσσερα κεφάλαια. Θα γράψουμε εκ νέου τα κεφάλαια 1 έως 4. Αυτό όμως που φοβόμαστε είναι ότι το κείμενο θα παγώσει. Οι εξελίξεις θα παγώσουν. Βλέπουμε γενικά μια τάση προσυνένεση συνένεση από τα κράτη-μέλη. Ήδη την προηγούμενη εβδομάδα και αυτή την εβδομάδα στην Κορεπέρ συζητούμε ορισμένα από αυτά τα θέματα για να δούμε αν μπορούμε να αποκλείσουμε κάποια επιμέρους συζητήματα. Την παρασμένη εβδομάδα συζητήσαμε το πεδίο εφαρμογή, για παράδειγμα. Επίσης θα συζητήσουμε τον ε, ορισμό της συνένεσης και της ελευθερίας του λόγου και της έκφρασης. Να σας υπενθυμίσω ότι στο τέλος του περασμένου Συμβουλίου ο υπουργό μου είπε ότι είναι πολύ σημαντικό να προχωρήσουμε με προσοχή και στο τέλος της όλης διαδικασίας να έχουμε σχεδιάσει μέσα τα οποία μπορούν να αντιμετωπίσουν και να διαχειριστούν όλο αυτό το νομοθετικό πακέτο. Όσον αφορά τον δημόσιο τομέα τώρα, οι αρμόδιοι υπουργοί κατέστησαν σαφές ότι καταρχά χρειάζεται περισσότερη ευελιξία ε, στον δημόσιο τομέα στα πλαίσια του κανονισμού αυτό όμω δεν θα ολοκληρωθεί κάτω από την Ιρλανδική Προεδρία, αλλά από την επόμενη. Ευχαριστούμε πολύ. Δεν ακούγεται και ιδιαίτερα θετικό αυτό που μας λέτε, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν βλέπω κάποιον από την υπηρεσία EDPS προστασίας ε, δεδομένων. Θα επιστρέψω λοιπόν στον εισηγητή. Κύριε Άλμπρεχτ, ευχαριστώ πολύ. ορισμένα σύντομα σχόλια πάνω στις ανησυχίες των μελών. Κύριε Βάντεκαμπ, για όλα αυτά τα σημεία που αναφέρετε μπορώ να σας πω ότι τα επεξεργαζόμαστε. Ήδη. Ιδιαίτερα όσον αφορά την έρευνα, προσπαθούμε μαζί να βρούμε μία λύση η οποία θα απαντά στους προβληματισμούς που διατυπώθηκαν πιστεύω πως είμαστε, απέχουμε πολύ λίγο από το να βρούμε μια συμβιβαστική λύση. Ήδη έχουμε προχωρήσει αρκετά. Και έχω την αίσθηση ότι αυτοί οι συμβιβασμοί, αυτές οι συμβιβαστικές τροπολογίες θα αντιμετωπίσουν αυτούς τους προβληματισμούς σας. Τώρα όσον αφορά το δικαίωμα κάποιου να λησμονηθεί, το right to be forgotten, έχουν προταθεί ορισμένε διατάξει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Προσπαθούμε αυτέ να τι εναρμονίσουμε. Φυσικά πιστεύουμε ότι αυτές οι πρόσθετες διατάξεις για το ψηφιακό περιβάλλον συγκεκριμένα, αλλά και γενικά θα αντιμετωπίσουν τις συνέπειες της επεξεργασίας των δεδομένων, πιστεύω πως θα μπορέσουμε να βρούμε λύση η οποία θα βασίζεται στην πρότασή μου. Τώρα, κυρία Λόπες, μπορώ να σας πω ότι όσον αφορά την συγκατάθεση και την δυνατότητα απόσυρσης της συγκατάθεσης, ήδη έχουμε βρει μια διατύπωση έτσι ώστε να διασφαλίζεται και να ενισχύεται το δικαίωμα αυτό. Και όσον αφορά τις αρμοδιότητες ανάμεσα στις αρχές. Εδώ θα ήθελα να σας παραπέμψω και στην πρόταση της έκθεσής μου, σύμφωνα με την οποία θα πρέπει να υπάρχει μία, η λύση μίας στάσης, μία λύση και επίσης θα πρέπει να είναι καθήκον αυτής της υπηρεσίας, αυτού του οργανισμού να συντονίζει την επιβολή του νόμου και να συμφωνήσουμε σε έναν σε μια κοινή ερμηνεία που θα υιοθετείται από όλες τις αρμόδιες αρχές και από εκείνες που θα εκπροσωπούν τους πολίτες. Είναι βέβαια πολύ σημαντικό το ζήτημα, το τονίσατε και εσείς οι ίδιοι εξάλλου, πολύ σημαντικό για τους πολίτες. Και το να υπάρχουν πολλέ ε, διαφορετικέ γλώσσε ή πολλέ διαφορετικέ αρμόδιες αρχέ ανά κράτος είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε να δημιουργήσει προβλήματα. Τώρα, κύριε Εντφέλτ, ακολουθούμε αυτήν την προσέγγιση δέσμης ως κοινοβούλιο, να σας απαντήσω. Θέλουμε να κάνουμε παράλληλες διαπραγματεύσεις και για τον κανονισμό και για την οδηγία. Και το πεδίο εφαρμογή του κανονισμού θα πρέπει να περιοριστεί, ιδιαίτερα όσον αφορά τις δημόσιες αρχές, στα συμπεράσματα του ψηφίσματος ε, του 2011, της έκθεσης ΦΟΣ δηλαδή, ότι δηλαδή εμείς θέλουμε να υπάρχει ένα ενιαίο όργανο, μια ισχυρή νομική βάση, επιβολή του νόμου, μπορούμε να το δεχτούμε αυτό από την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν θα πρέπει όμως να αλλάξει παραπάνω. Τώρα κάτι άλλο που θα ήθελα να θίξω διότι πολλές ε, ομάδες με ρώτησαν σχετικά για τα δημόσια αρχεία, για το πώς επεξεργάζονται αυτά τα προσωπικά δεδομένα. Εδώ θα ήθελα να πω ξεκάθαρα ότι όλες οι κοινοβουλευτικές ομάδες και οι εκπρόσωποι τους συμφώνησαν στο ότι οι δυνατότητες που έχουν, ε, οι δυνατότητες ύπαρξης αυτών των δημόσιων αρχείων θα πρέπει να μειωθούν και από, από εκεί που είναι σήμερα θα πρέπει να αλλάξει η νομοθεσία έτσι ώστε να, γίνεται, να γίνει δυνατή και σαφέστερη η λειτουργία τους μέσω του κανονισμού. Και φυσικά τα κράτη-μέλη, είτε με κοινοτική είτε με εθνική νομοθεσία, θα πρέπει να διευκρινίσουν και να δώσουν πλαίσιο στον, στις αρμοδιότητες των όσων επεξεργάζονται και συλλέγουν αυτά τα δεδομένα. Πάρα πολλές ανησυχίες διατυπώθηκαν ιδιαίτερα ως προς αυτό το σημείο και πιστεύω πως θα μπορέσουμε να συμφωνήσουμε σε ένα κείμενο. Πραγματικά λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη όλους αυτούς τους προβληματισμούς στις συζητήσεις μας. Θέλουμε, τονίζω, να προχωρήσουμε με μια ευρεία συνένεση και να το κάνουμε αυτό γρήγορα. Διότι πραγματικά βλέπουμε εμείς εδώ στο Κοινοβούλιο ότι έχουμε τη δυνατότητα να Έχουμε στα χέρια μας ένα όργανο που θα μας δώσει σαφήνεια, νομική σαφήνεια και ένα πλαίσιο για όλους. Τώρα όσον αφορά τις τεχνικές ε, δυνατότητες ανταλλαγής δεδομένων σε διασυνοριακή βάση, πιστεύω πως τώρα έχει έρθει η ώρα να προχωρήσουμε με τον κανονισμό, με την οδηγία και να προσπαθήσουμε να οριστικοποιήσουμε τις θέσεις μας εδώ στο Κοινοβούλιο πριν το καλοκαίρι και πραγματικά χρειάζεται προσπάθεια από όλους μας, από όλα τα κράτη-μέλη και από την Ιρλανδική Προεδρία έτσι ώστε αμέσως μετά το καλοκαίρι να αρχίσουμε τις διαπραγματεύσεις. Πιστεύω πως είναι κοινό μας στόχος και κοινό συμφέρον να ολοκληρώσουμε τους φακελούς αυτούς πριν τις επόμενες εκλογές. Οι πολίτες θέλουν να δουν αποτελέσματα και εμείς πρέπει να καταβάλουμε προσπάθειες. Καταβάλουμε ήδη προσπάθειες και η Ιρλανδική Προεδρία. Το βλέπουμε αυτό. Πρέπει λοιπόν να συνεργαστούμε από κοινού έτσι ώστε να ολοκληρώσουμε αυτή τη διαδικασία και να έχουμε καλά αποτελέσματα. Και είμαι πεπισμένος ότι θα τα έχουμε. Ευχαριστώ. Ωραία. Φτάνουμε στο τελευταίο σημείο της σημερινής διάταξης σήμερα, το οποίο θα είναι λίγαν σύντομο για τη στρατηγική ασφάλειας του κυβερνοχώρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. έχω τώρα μία νέα έκδοση του σημειώματος ενημέρωσης. Ε, okay. well, it's going to be even shorter, so that's good. Ακόμα σύντομότερο θα είναι αυτό το θέμα. Η στρατηγική ασφάλειας του κυβερνοχώρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης εγκρίθηκε από την Επιτροπή σε 7 Φεβρουαρίου η ανακοίνωση και η ΙΜΚΟ, η Επιτροπή ΙΜΚΟ έχει ε, προετοιμάσει ένα προσχέδιο έκθεσης. Ο κύριος Σφάπ είναι ο εισηγητής, αλλά δεν είναι διαθέσιμο το κείμενο, γι' αυτό προτείνω να αναβάλουμε τη συζήτηση. Θα λάβετε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο την πρόταση. Στις 14 Μαΐου είναι, έχει οριστεί η προθεσμία για υποβολή τροπολογιών και στις 29 και 30 Μαΐου θα ψηφίσουμε στη ΛΥΜΠΕ και θα υποβάλουμε και τροπολογίες. Και βλέπω ότι όλοι ήδη φεύγετε προς το Place de για να ε, μπορέσετε να εποφαληθείτε από τις ε, πρώτες, μία από τις πρώτες ανοιξιάτικες μέρες. Λύεται η συνεδρίαση.